Okay, can we start the meeting? Okay, thank you. Uh, uh thank you for being here. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που ήρθατε και ξεκινάμε πρώτα-πρώτα έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε τους διευθυντές ε, στα πλαίσια της Αρμοδιότητας Επιτροπής. Επίσης έχουμε την έκθεση του Eurofound για σύνθεση και ευημερία των οικογενειών. Συμφωνείτε για την ημερήσια διάταξη. Ωραία. Ανακοινώσει της Πρόεδρου. Έχουμε σε όλες τις γλώσσες ε, διερμηνία και όποιος ψάχνει τη γλώσσα του κοιτάξτε στον φωτεινό πίνακα το κατάλληλο νούμερο για σας και όπως έχουμε τις ανταλλήγα από τους διευθυντές αρμοδιότητά μα, ε, Πέντε είναι αυτές οι υπηρεσίε και οργανισμοί σε σχέση με τα θέματά μα Εκείνοι παραδοσιακά προσκαλούνται ε, στις αρχέ κάθε χρόνου στην Επιτροπή μας για να παρουσιάσουν το έργο του οργανισμού τους. Ε, ίσως ο Τζόρντι Κουρέλ είναι καινούριο και δεν το ξέρει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης οι υπόλοιποι όμω ε, τα ξέρετε, ε, όπως ο κύριος ε, Ζίμπελ, ο εκτελεστικό διευθυντής του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Επίσης είναι ο γνώριμο και ο Χουάν Μενέντε Βαλντέ, ο εκτελεστικό διευθυντής του Eurofound. Επίσης τα γνωρίζει και τη γνωρίζουμε την Κρίστα Σέντλατζεκ, την εκτελεστική διευθύντρια του ΩΣΑ. Και επίσης παλαιός γνωστός και ο διευθυντής του ETF, ο Τσέζαρε Ονεστίνη. Με αυτή την ευκαιρία να σας τονίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η οργανισμή και η για το έργο της Επιτροπής μας. Από πλευρά τη Επιτροπή, ευχαριστούμε για τη συνεργασία στο παρελθόν και συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, έχουμε καλέσει και κάποιους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με αυτές τις ε, υπηρεσίες. Και θα τους δώσουμε αργότερα τον λόγο στον κύριο Μπέκερ για το Σέντεφοπ, στην κυρία Λόπε Φοντανιέ για την Eurofund, για τον κύριο Μίσιτς για την EU όσα Θέρκας και Μπάουρ για το ETF και Κρέμερ για τον ELA. Καλώ ορίσατε όλοι. Πρώτη φορά μας επισκέπτεστε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ξεκινούμε και να δώσουμε το λόγο στους διευθυντές. Έχετε περί τα 10 λεπτά έκαστος για την παρουσίαση σας. Και ο εξαριστερός μου θα έχει το ο κύριος Ζίμπελ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές. Ευχαριστούμε μας καλέσατε και πάλι να σας πω για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, για τις ε, αξίες, τους στόχους, τις πολιτικές μας, τι κάνουμε για αυτές, ε, στρατηγικές ε, κινήσεις και ευχαρίστως να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Το 75 συγκροτηθήκε η υπηρεσία μας, όπως βλέπετε εδώ στην διαφάνεια, ούτω ώστε να προωθήσουμε τα θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης. Συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπειρογνώμονες, συγγνώμη με όλους τους και συνεργαζόμαστε βέβαια και με άλλες ε, υπηρεσίες, με τα κράτη-μέλη ε, και αυτά όλα σε σχέση με την διαδικασία της Κοπενχάγης Και έχουμε τον ορίζοντα πολιτικής του 2020, αλλά το 2007 αναβαθμιστήκαμε όσον αφορά τον ρόλο μας για την πλαίσιωση των πολιτικών. Και γνωριζόμαστε ως ε, άργος των νέων όσον αφορά επίσης τις δεξιότητες και τις ικανότητες, τις επαγγελματικές και ε, επίσης όσον αφορά την διάδοση των γνώσεων για όλους τους εμπλεκόμενους. Έχουμε το καταστατικό μας, το ιδρυτικό, το οποίο έχει τροποποιηθεί το 2019. Έχουμε νέο καταστατικό και τώρα έχουμε επίσημη αναγνώριση για κάποιες λειτουργίες που έχουν ε, γίνει εδώ και κάποιο καιρό όσον αφορά την ε, αγορά απασχόληση και τις δεξιότητες. Οπότε, προσπαθούμε έτσι να κάνουμε ό,τι πρέπει με κάποιο τρόπο αξιόπιστο να λάβουμε υπόψη κάποια στοιχεία, τις νέες γνώσεις, να παρακολουθήσουμε τις πολιτικές και όπως είπαμε να είμαστε κάτι σαν διαμεσολαβητής ε, στις σχετικές γνώσεις και πληροφορίες μεταξύ κρατών μελών και των εμπλεκομένων. Επίσης ε, είχαμε τη δέξη της Κοπενχάγης, σας το είπα, ε, αυτά φέρνουν το παρελθόν, αλλά για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εδώ υπάρχει το θέμα το ε, έργο μας με ορίζοντα το 2030. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη υπάρχει κάποια πρόταση που έχει εγκριθεί από την Συμβουλευτική Επιτροπή για την ε, κατάρτιση, το ECVT και έχουμε μόλις τη νέα ε, ε, πολιτική. Τώρα έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πολύ σημαντικό αυτό και στα πλαίσια της νέας πράσινης συμφωνίας που ε, μας οδηγεί σε, σε πράσινη παιδεία, πράσινη εκπαίδευση, πράσινη απασχόληση. Επίσης ε, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, νέες δεξιότητες, την, ε, το εγγυητικό μέσο πολιτική των για τους νέους. Επίσης έχουμε και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και αυτό είναι πέραν όλων των άλλων στόχων μας που βέβαια είναι αυτονόητη στα πλαίσια της κατάρτισης. Ε, τώρα, βλέπετε τώρα τους στρατηγικούς λειτουργία ε, λειτουργίας ε, για το πώς διαμορφώνουμε την κατάρτιση και προσανατολισμό, πώς γίνεται η αξιοποίηση, η χειραφέτηση και ενημέρωση. Επίσης, θα πρέπει να σας πω και κάποια στοιχεία. Ελπίζω ότι από αυτά τα στοιχεία, που βέβαια δεν είναι αυτονόητο, να δείτε ε, ποια είναι τα αποτελέσματα του έργου μας. Αλλά βέβαια εμείς ε, ως ε, οργανισμός πρέπει αυτό να το καταγράψουμε. Νομίζω ότι είναι αυτά τα στοιχεία εντυπωσιακά και βέβαια σας παραπέμπω και στην μαρτυρία των τριών θεσμικών οργάνων αλλά και των κοινωνικών εταίρων και ε, διεθνών φορέων που ακριβώς είναι μάρτυρες του έργου μας ο ΑΕΛΟ, η UNESCO τώρα. Όσον αφορά τον προπολογισμό και την εκτέλεσή του, βλέπετε εδώ τα στοιχεία και θέλουμε εσείς που είστε αρχή του προπολογισμού να μας ε, βοηθήσετε και έτσι να συνεχίσουμε το έργο μας. Παρ' όλα αυτά η πορεία μας η καλή ε, φρενάρισε λίγο πριν τα Χριστούγεννα επειδή είχαμε περικοπή 300 εκατομμυρίων. Αυτό βέβαια δεν γίνεται κάθε μέρα. Βλέπουμε τώρα τι άλλο για, τα, για το ε, έργο μας. Βλέπετε και δίπλα στην πόρτα ένα, αυτό το, το, το, το έντυπο, το ενημερωτικό είναι ένα σημείωμα και έχει σχέση με αυτά, αυτά που τα βλέπετε εδώ δεξιά στη διαφάνεια για τις δημοσιεύσεις μας. Περιγράφουν τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν, ε, διάφορες ε, δημοσιεύσεις. Βλέπουμε και ωραίους τίτλους, ε, δεξιο, προγνωστικά δεξιοτήτων, ευρωπαϊκές δεξιότητες κλπ. Όλα αυτά είναι το έργο μας που δια, διαπνέει αυτές όλες τις ε, δημοσιεύσεις και όπως βλέπετε στο δεξιό τμήμα της διαφάνειας όλο ένα και περισσότερο προσπαθούμε να δώσουμε και ιντερνετικά ε, κάποια στοιχεία. Εδώ έχω, βλέπετε 12 εικονίδια στα αριστερά. Είναι οι εκδόσεις μας το 19 και το 20, Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων. Ε, είναι προσέγγισή μας για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης και προσανατολισμό Επίσης υπάρχει εδώ ένα εργαλείο για την μαθητεία ε, δεξιότητες, ανάλυση διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης ή κενών θέσεων απασχόλησης και το 2018 αναπτύξαμε αυτό το, το εργαλείο προγνωστικών ε, και άλλου είδους μέσα προσανατολισμού. Έτσι προσπαθούμε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στο υλικό που έχουμε και σας ζητώ αυτά που σας λέω να τα δοκιμάσετε. Πιέζει χρόνος και προχωρούμε ε, όχι σε άλλα αποτελέσματα που θα ήθελα, αλλά όποιο θέλει να του τα πω διμερός. Επίσης, εδώ έχουμε αναλύσει τις τάσεις ε, της ζήτησης να αγορά εργασίας, κάποια δημογραφικά στοιχεία επίσης έχουμε, αλλά και αυτά τα παραλείπω, αλλά προτιμώ να σας πω τι γίνεται όσον αφορά την έλλειψη σε επίπεδο δεξιοτήτων που έτσι μας κολοβώνουν ε, τις δυνατότητες ως Ένωση και να δείτε εδώ τι λέμε για αυτές τις ε, ελλείψεις. Θεωρούμε ότι αυτό θα αυξήσει το κόστος εργασίας. Έχουμε εδώ την διαρθρωτική ανεργία, έχουμε την επιβράδυνση της ε, ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι βέβαια και μακρόπνοα αρνητικά για τις επενδύσεις. Βλέπετε δεξιά ακριβώς τι γίνεται όσον αφορά αυτές τις ελλείψεις δεξιοτήτων, τι γίνεται με τις εταιρείες καινοτομίας, τις αναπτυσσόμενες εταιρείες, ε, οικοδομικές και αυτές που έχουν δυσκολία ε, πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά. Δεν έχουμε χρόνο, λέει ο μιλητής και μιλάει ένα και πιο γρήγορα και γι' αυτό είναι δύσκολο να μεταφραστεί πλήρως. Α, τώρα, τώρα πηδήξαμε 5-6 διαφάνειες και ε, έχουμε τώρα αυτήν την ε, μελέτη Crowd Learn. Και βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται 19 Μαρτίου. Έχουμε μια, μια εκδήλωση για να δούμε τι γίνεται με την οικονομία της πλατφόρμας και το Crowdwork. Επίσης βλέπετε τώρα αυτόν τον υπέροχο ναό για να ολοκληρώσω την ανάλυση μας όσον αφορά τις κενές θέσεις εργασίας. Βλέπουμε που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στην ε, ανατομέα. Βλέπουμε ε, τι πρέπει να κάνουν ε, οι Ευρωπαίοι, δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και άλλες οριζόντιες και έτσι διαμορφώνονται τα συστήματα κατάρτισης και προσανατολισμού, χρηματοδότηση, πρόσβαση. Έχουμε τη μετάβαση, την πράσινη, την ε, ε, ψηφιακή. Όλα αυτά τα προσεγγίζουμε όλα μαζί γιατί είναι αλληλένδετα οπότε το κλειδί για τη δουλειά μας είναι αυτά τα εργαλεία, η χρηματοδότηση και ευρεία δυνατότητα πρόσβασης. Στα αριστερά βλέπετε αυτό το βελάκι που λέει για την ε, για την ανάπτυξη της πολιτικής εφαρμογής και για δεξιά βλέπετε την συνεισφορά στη διαμόρφωση αυτής. Εδώ βλέπετε τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου μας το 20. Τέλος πάντων για το 20. Ε, ευφία σχετικά με τις ε, δεξιότητες, ανάπτυξη δεξιοτήτων και παρακολούθηση των ε, εξελίξεων όσον αφορά κατάρτιση και προσανατολισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που με ακούσατε και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Αργότερα θα έχουμε ένα γύρο απαντήσεων. Ο Χουάν Μέντεθ Βαλντές όμως τώρα είναι ο επόμενος. Παίρνει τη σκητάλη να μας μιλήσει. Για πού? Α, για το Eurofund, μάλιστα. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Επιτροπή σας. Ορισμένοι από εσάς ήταν βουλευτές και στην προηγούμενη θητεία. Και θέλω να σας ευχαριστώ ιδίω γιατί είναι η τελευταία φορά που έρχομαι σε αυτή την ε, ανταλλαγή απόψεων για την παρουσίαση των ετήσιων προγραμμάτων στα τέλη του έτους λίγη η θητεία μου, τέλη Δεκεμβρίου του 2020. Ελπίζω πάντως να έχω χρόνο να συμμετέχω σε άλλες συζητήσεις, όχι πάντως σε αυτήν την άσκηση. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη στήριξη που παρέχετε όλα αυτά τα χρόνια στον οργανισμό μας. Η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά αλλαγών, δεν θα επαναλάβω τα προφανή, δηλαδή η αλλαγή του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν, αλλά και εμείς ε, είχαμε μια νέα ε, αδερφή υπηρεσία την αρχή για την εργασία. Έχουμε επίση ε, την εξωτερική αξιολόγηση που πρέπει να δοθεί συνέχεια και το σημαντικότερο ολοκληρώνουμε ήδη από φέτος το τρέχον πολιετές. Το προτελευταίο ολοκληρώθηκε πέρσι και φέτος άρχισε εφαρμογή του τελευταίου κύκλου. Στον κύκλο αυτό έχουμε τους τέσσερις πυλώνες όπως τους αποκαλούμε που είναι βασική τόμη δραστηριοτήτων που άπτονται των συνθήκων εργασία και τη βιώσιμη εργασία, ποιότητα εργασία, προποθέσει, συνθήκε για να μπορεί κανεί να εργάζεται περισσότερο αν αυτό απαιτούν δημογραφικέ αλλαγέ. Δεύτερο πυλώνα είναι οι εργασιακέ σχέσει, διότι οι κοινωνικοί εταίροι ε, διαμορφώνουν και τι συνθήκε εργασία ε, από κοινού με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης έχουμε τις αλλαγές ε, στην αγορά εργασία, αναδιορθώσεις κτλ. Και τέταρτος πυλώνας ποιότητα ζωής και δημόσιας υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, ε, των τεσσάρων αυτών στρατηγικών προτεραιότητων έχουμε και δύο εγκάρσεις προτεραιότητες. Μια αφορά την ψηφιοποίηση πώς την επεξεργαζόμαστε και πώς αυτή επηρεάζει ιδίω στον κόσμο της απασχόλησης. Ε, έχουμε κάνει πολλή δουλειά όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτό το τομέα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι η παρακολούθηση της σύγκλησης στην Ευρώπη. θα σας αναφέρω όλα τα αποτελέσματα ή όλο το έργο το οποίο θα εκτελέσουμε. Μπορείτε να τα διαβάσετε στα επίσημα έγγραφα του Eurofound. Αλλά κάποιες βασικές ε, γραμμές, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τον πρώτο στρατηγικό πυλώνα, μαζί με τον Οργανισμό Εργασίας, το ILO, έχουμε μια κοινή έκθεση δημοσιεύση, καλύπτοντα 41 χρόνες, ε, χώρες και 1,5 δισεκατομμύρια εργαζομένους ανά τον κόσμο για να δούμε ποια είναι η ποιότητα της απασχόλησης. Είπα Νότια Κορέα, κάποιος πόλει της Κίνας και κάποιες λατινοαμερικανικές χώρες μεταξύ άλλων. Δεύτερη εστίαση, δεν θα εξαντλήσω όλα τα θέματα, ήταν η συμφιλίωση εργασιακού και ιδιωτικού βίου. Για να δούμε επίσης τι γίνεται με τους πατέρες, τις μητέρες, ε, τι προτιμούν να κάνουν, γονική άδεια, εργασία γιατί είχαμε και την οδηγία για την ε, συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και για τους φροντιστές και για τους γονείς και θέλαμε να δούμε πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις. Επίσης βλέπετε τι δημοσιεύσαμε την κοινή εκθέση για την απασχόληση του 2020. Καλύπτει τις θέσεις εργασίας ποιότητας αλλά και άλλα θέματα. Επίση, εστιάσαμε σε άλλες παρουσιάσεις μα στο ωράριο εργασίας, στο χρόνο εργασίας. Είδαμε επίσης και τα θέματα της οροπία μεταξύ ε, εργασιακού και οικογενειακού και θέματα φύλου ε, επί ρουμαϊκή προεδρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει το 2020, θα έχουμε 40.000 συνεντεύξει ε, με εργαζομένου από όλε τι χώρε. Περιλαμβάνω εδώ ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο, που εξακολουθεί να είναι μέλο μια επιτόπου εργασία. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία για το Ηνωμένο Βασίλειο πριν συμφωνήσει, πριν πράξη συμφωνία για τον Brexit. Εστιάζοντας και εδώ στην ποιότητα. Έχουμε επίσης μια εμβληματική έκθεση που θα τονίσουμε διάφορα θέματα. Δεν θέλω να τα αναφέρω όλα για να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές και οι προκλήσεις. Επίσης θα κάνουμε κάποια δουλειά για την τηλεεργασία και το δικαίωμα στην αποσύνδεση, που φαντάζομαι ότι θα το συζητήσετε εδώ. Δεύτερος πυλώνας, εργασιακές σχέσεις. Έχουμε κάνει πολλά εδώ. Αυτό όμως που μας απασχόλησε περισσότερο ήταν κατώτατη μισθή. Είδαμε επικαιροποιημένα στοιχεία, ε, πώς εξελίσσονται καθάριστη μισθή, τι μπαίνει στην τσέπη των Ευρωπαίων εργαζομένων τελικά και όλα αυτά τα στοιχεία τα αξιοποιήσαμε με την έρευνά μας. Στη διαβούλευση για ένα έγγραφο που ξεκίνησε από την Κομισιόν το Γενάρη, στις 14 μήνες. Και ένα δεύτερο είναι η αντιπροσωπευτικό των κοινωνιτέρων στον τομεακό διάλογο. Επίσης θα έχουμε φλάξιπ, εμβληματική έκθεση, αλλά κυρίως για τους κατώτους μισθούς. Καλύψαμε και άλλους τομείς στην κοινή έκθεση για την απασχόληση και στις διαβουλεύσεις για τους κατώτους μισθούς. 2020 θα συνεχίσουμε. Έχουμε μία έκθεση εμβληματική που θα ε, συνδυάζει διάφορα πορίσματα στον τομέα αυτό το κάτω μισθών. Θα στηρίξουμε τις συζητήσεις για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τη δημιουργία υποδομών και ικανοτήτων. Ικανοτήτων δε για τους κοινωνικούς εταίρους. Και έχουμε και τις επερχόμενες συζητήσεις. Θα έχουμε διαφάνεια μισθών και διάσταση του φύλου. Στο χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, μερικά θέματα που θα καλύψουμε. Εσείς ε, λάβατε μία παρουσίαση για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις πρόσφατα και Υπάρχει και συζήτηση η οποία θα οργανωθεί από τους Αλισσάς και Δημοκράτες το Φεβρουάριο για τους ε, κατώτατους μισθούς. Τώρα, τρίτος πυλώνας, αλλαγές στην αγορά εργασίας. Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα εδώ, μια ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις. Από κοινού με τους Αντεφόπ και το ΆΙΖΑ. Πολύ καλή συνεργασία, στο καλύτερο παράδειγμα συνεργασία μεταξύ των τελεστικών οργανισμών. Και οικονομικά μοιραζόμαστε τον προπολογισμό αλλά και καλύπτουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα. Πάνω από 30.000 εταιρείε. Ε, τα αποτελέσματα θα τα πάρετε φέτος και θα δημοσιοποιηθούν γενικά. Και με το ΙΖΑ, το Ινστιτούτο Οικονομικών, στον τομέα της εργασίας. Μας βοήθησε. Επίσης, ε, το μέλλον ε, της μεταποίησης ήταν ένα άλλο θέμα. Είδαμε κάποιες εκτιμήσεις και κάποια σενάρια με πιο επιτυχημένο το σενάριο την υλοποίηση των στόχων της Φωνής των Παρισίων. Και επίσης έχουμε τα μέτρα αυτά που θα οδηγήσουν σε ε, μια ποσοστία μονάδα ανάπτυξης και 0,5% ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Βέβαια, ανάλογα με του τομεί και τι χώρε, κάπου μπορεί να έχουμε απώλειες σε θέσει εργασία, κάπου μπορούμε να έχουμε αύξηση. Είδαμε επίση τον διαχωρισμό τη αγορά-εργασία και συνεχίζουμε τη δουλειά μα, βέβαια, για τι ε, δομικέ αλλαγέ στην αγορά-εργασία. Πολλέ ε, ε άλλε συνεισφορέ ε, στο policy uptake στην έκθεση για την απασχόληση και για την εξελίξει τη κοινωνική τομέα τη απασχόλησης έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το κλίμα και κάποιες άλλες αναλύσεις. ελλείψη εργατικού δυναμικού κτλ. Και θα βοηθηθούμε και από τα αποτελέσματα άλλων οργανισμών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο να πάω στην ποιότητα ζωή, δημόσιε υπηρεσίε. Εδώ είχαμε μια έκθεση εμβληματική και θα ακούσετε και τα σχετικά με τη σύνθεση και την ευημερία των νοικοκυριών αργότερα στη σημερινή σα συνεδρίαση. Κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Παγκόσμιο Οργάνωση υγεία. ανέλησε τα στοιχεία του IQS της Ένωσης, της ε, έρευνας της Ένωσης για την ε, ποιότητα της υγείας. Και γιατί υπάρχουν διαφορές. Το 2020 τι θα κάνουμε. Θα ξαναδούμε την κατάσταση των ανθρώπων αυτών που ούτε εκπαιδεύονται, ούτε ε, είναι ασκούμενοι, ούτε έχουν εργασία, οι νίτς, οι λεγόμενοι και διάφορα άλλα. Και η εργασιακή φτώχεια θα μας απασχολήσει. Ψηφιακό, ψηφιακή εποχή θα εστιάσουμε στις πλατφόρμες. Θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις. Νομίζω θα γίνει ένα γεύμα ε, το οποίο θα γίνει το Μάρτιο με ευρωβουλευτές και επίσης θα δούμε και διάφορα άλλα σενάρια σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτή τις πλατφόρμες και το έργο τους. Και τέλος, ε, η σύγκληση. Έχουμε και καλά και κακά Είδατε ότι είχαμε το 2019 διάφορες παρουσιάσεις, συμμετείχαμε στις ε, συνεδριάσεις ΕΜΚΟ και SPC. Πάρα πολύ γρήγορα κάποια αποτελέσματα. 95% είναι τα ικανοποίηση, τα ποσοστά ικανοποίηση στην έρευνα αυτή που κάναμε για την κάμψη των χρηστών. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα, 94% ικανοποίηση για την αξιοπιστία των δεδομένων, για το πόσο σχετίζονται αυτά που κάνουμε με το θεματολόγιο και 82% ικανοποίηση σε ό,τι αφορά για άλλους. Και ποιοι είναι βασικοί δείκτες επιδόσεων. 160 έγγραφα χρησιμοποιούν τα δικά μας πορίσματα και documents, βασικά ε, έγγραφα, Βασικοί πελάτες, Κομισιόν και Κοινοβούλιο, 210 συμμετοχές εξωτερικών σε εκδηλώσεις, χιλιάδες ε, ε, μεταφορτώσεις εγγράφων και πολλά άλλα. Συνεργαζόμαστε με άλλους οργανισμούς, αλλά δεν έχω χρόνο για να τα πω με αστρονομική ταχύτητα όπως τα λέω μέχρι τώρα, οπότε θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα. Θα ξεκινήσουμε με τον ΕΛΑ που είναι αυτή η αρχή για την ε, εργασία και έχουμε ξεκινήσει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καθότι είμαστε στην προετοιμασία του νέου κύκλου και θα πρέπει να δούμε τον προτέρων που θα εστιάσουμε. Και δεν θα εστιάσουμε μόνο στην ψηφιοποίηση, αλλά και στην ε, μετάβαση και στην κλιματική αλλαγή. Και όταν μιλάμε για τη σύγκληση, δεν θέλουμε να περιοριστούμε στην κοινωνική σύγκληση, αλλά να δώσουμε προσοχή και στο θέμα, στον, στην έννοια τη κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ ε, πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή η τελευταία σας παρουσίαση υπό την ιδιότητα αυτή. Ε, θα έχουμε τη δυνατότητα ε, να ξανασυστήσουμε κατά τη διάρκεια του έτους. Δεν νομίζω καν ότι έχουμε στείλει ακόμη την πρόσκληση για γεύμα εργασίας στις 19 Μαρτίου. Πάντως όσοι είστε παρόντες μπορείτε να σημειώσετε την ημερομηνία αυτή διότι θα οργανώσουμε τη συνάντηση αυτή ε, σε συνεργασία με τους δικούς μας οργανισμούς εντός εισαγωγικών. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Κρίστα Σέκ για την τρίτη παρουσίαση που είναι ε, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία Συνεργασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλημέρα και στους Ευρωβουλευτέ της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια επισκόπηση των όσων συνέβησαν το 2019 και να κάνω κάποιες προβλέψεις για το 2020. Είχαμε ένα έτος συναρπαστικό και επιτυχέ. Ε, γιορτάσαμε την 23η επέτειό μας, ε, το οποίο σημαίνει ότι, ε, ότι συμβάλλουμε εδώ και 25 χρόνια ε, στην ευελτίωση των συνθήκων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επιτυχία. Συγκεντρώνουμε, αναλύουμε και ε, δημοσιεύουμε πληροφορίες και χρησιμοποιούμε επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας ε, για την ε, ασφάλεια και την υγεία στην ε, εργασία. Οργανώσαμε την μεγαλύτερη εκστρατεία μας. Η τελευταία ολοκληρώθηκε τέλη του προηγούμενου έτους για τις επικίνδυνες ουσίες. Πολύ σημαντικό θέμα και τον Οκτώβριο κατά τη διάρκεια ε, της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για μειοσκελετικές διαταραχές θα, ξεκινήσουμε επίσης νέα εκστρατεία. Αναφέρθηκε ήδη ο κανονισμός ίδρυσής μας από το 2009. Ε, Εργαζόμαστε με βάση αυτόν τον κανονισμό και είχαμε εναρμόνιση ε, με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Αυτή ήταν μια θετική εξέλιξη και θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα το οποίο συμπεριλήφθηκε στον ιδρυτικό κανονισμό. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ήταν ο κρίκος που έλειπε τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχουμε ανεξάρτητο ε, επόπτη για την ασφάλεια και την υγεία συνεργασία ε, στις συνεδριάσεις ε, του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως ήδη αναφέρθηκε ο κύριος Φλακμίτσης και, και ήδη συμμετείχε την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, συνεδρίαση του Διευθυντικού Συμβουλίου. Ήταν θετική η πρώτη μας συζήτηση και είμαι πεπισμένη ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και ε, πιο στενή συνεργασία με ε, το, την Επιτροπή Απασχόλησης ε, και το Κοινοβούλιο γενικά. Αναφέρθηκαν ήδη διάφορες αλλαγές, το, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, ο Ιδρυτικός Κανονισμός. Υπάρχουν όμως ε, πολλές ενδείξεις ε, που δείχνουν ε, ότι η ασφάλεια και η υγεία συνεργασία συνεχίζουν να είναι σημαντικός τομέας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με ένα νέο βιντεομήνυμα στην ιστοσελίδα μας που ετοίμασε το γραφείο του, του νέου επιτρόπου του κυρίου Σμιτ ο οποίος ε, μεταφέρει το πολύ σημαντικό μήνυμα ότι η ασφάλεια και η υγεία συνεργασία παραμένουν ε, ε, σημαντικό θέμα για την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέε μορφέ εργασία, οι νέε τεχνολογίε. Αποτελεί προτεραιότητα οι εργαζόμενοι να είναι ασφαλείς και υγιείς, όχι μόνο μέχρι την ημερομηνία συνταξιδότησής τους. Επίσης, εκδόθηκε έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, έχει να κάνει με τους ε, οργανισμούς απασχόλησης και δεν διαπιστώθηκε λόγος για σημαντικές αλλαγές στον ίδιο e όσα φυσικά. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει συστάσεις για καθέναν από τους οργανισμούς μας ε, και φυσικά θα λάβουμε υπόψη μας τις συστάσεις αυτές. Συζητάμε το πώς και πότε. Όπως ήδη είπα, το έτος 2019 ήταν έτος επιτυχιών. Είχαμε μεγάλη, ε, μεγάλο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επίσης είχαμε πολύ στενή συνεργασία, όλο και καλύτερη θεωρώ, με ε, τα εθνικά ε, σημεία εστίασης, τα εθνικά σημεία επαφής και όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου εργασιών μας, ε, αλλά και ε, όσον αφορά τους κοινωνικούς εταίρους και τη συνεισφορά τους στο έγγραφο εργασίας, στο πρόγραμμα εργασίας. Όσον αφορά τα αποτελέσματά μας για το 2019, γνωρίζετε ότι η βασική ομάδα στόχος μας είναι ε, αυτοί που χαράσουν πολιτική. Θέλουμε να τους υποβάλουμε συστάσεις, να τους δίνουμε μια εικόνα για την ασφάλεια και την υγεία συνεργασία στην Ευρώπη, ε, και φυσικά μας ενδιαφέρουν και οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, αυτή η ομάδα στόχος ε, συμπεριλαμβάνεται σε σχεδόν ό,τι και να κάνουμε, διότι πρέπει να προσαρμόσουμε τα εργαλεία μας στις ανάγκες τους. Δημοσιεύσαμε έρευνες προηγμένες καθώς και πληροφορίες σχετικά με ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Αυτό είναι ένα θέμα ε, συνεχούς ενδιαφέροντος, διότι βλέπουμε ότι οι εργασιακές ασθένειες αυξάνονται αντί μία από αυτές τις δημοσιεύσεις είχε να κάνει με τον καρκίνο και την καταπολέμησή του. Ε, το πώς επιστρέφουν οι εργαζόμενοι στην δουλειά μετά ε, από θεραπεία καρκίνου και ε, θα δούμε και άλλες δημοσιεύσεις ε, φέτος και του χρόνου, καθώς ε, και συστήματα παρατηρητών για τις εργασιακές ασθένειες. Κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ο, ο λόγος, η αναλογία κόστους-όφελους και συζητάμε ε, συγκεκριμένη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, το ILO και τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ε, πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά ατυχήματα, εργασιακά τραύματα και εργασιακές ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα Επίσης, ε, να επανέλθω στην εκστρατεία για ε, τον χώρο εργασίας, την υγεία στον χώρο εργασίας. Όπως σας είπα, οι εκστρατείες μας ε, έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα θέματα. Ολοκληρώθηκε η εκστρατεία μα για τι επικίνδυνε ουσίε και εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι ήταν η πιο επιτυχής μα εκστρατεία. διότι είχαμε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι παλαιότερα. Οι επικίνδυνε ουσίες και οι καρκινογενείς ουσίες, ιδιαίτερα που αποτελούν προτεραιότητα, είναι θέμα με το οποίο μπορέσαμε να συμβάλλουμε στο πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρία για τις καρκινογενείς ουσίες. Δημοσιεύσαμε επίσης ε, μια ευρία επισκόπηση πριν από ένα χρόνο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στον τομέα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη εργαλείων για τις επιχειρήσεις αυτές. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε βελτιώσει το επιγραμμικό εργαλείο για ε, την ε, ανάλυση κινδύνου ένα διαδραστικό εργαλείο. Θέλουμε έτσι να έρθουμε σε επαφή με περισσότερες ε, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο. Εξετάζουμε επίσης τους κοινωνικούς εταίρους, τους εμπειρογνώμονες στις οικοδομές και στη γεωργία, διότι αποτελούν ε, την ε, πλειοψηφία των ε, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επίσης, ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας για την έρευνα των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. 45.000 πρόσωπα είχαμε ως συνομιλητές και πιστεύουμε ότι έτσι έχουμε αξιόπιστα ε, στοιχεία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σε όλα τα κράτη-μέλη που μπορούμε να συγκρίνουμε με τα παλαιότερα στοιχεία που είχαμε. Ενδιαφέροντα νέα ευρήματα είναι η σημασία της ε, νομοθεσίας και για πρώτη φορά ρωτάμε πώς γίνεται αποδεκτή η ψηφιοποίηση σε επίπεδο επιχείρησης. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης ε, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και μάλιστα ένα βαρόμετρο για την υγεία και την εργασία στην εργασία σε όλη την Ευρώπη με βάση μια σειρά δικτών. Μπορεί κανείς ε, να δει τις ε, λεπτομέρειες ε, που αφορούν κάθε χώρα. Κοιτώντας τώρα το 2020, θα ήθελα να αναφέρω τρεις βασικές δραστηριότητες. Αυτήν για τις μειοσκελετικές διαταραχές που αποτελούν σημαντική αιτία για αναρωτικές άδειες και πρόορη συνταξιοδότηση το επόμενο 24μηνο, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο φέτος ε, θα διαρκέσει αυτή η εκστρατεία. Η ψηφιοποίηση επίσης αποτελεί σημαντική προτεραιότητά μας. Θα ξεκινήσουμε από μια επισκόπηση, έκθεση και διάφορες δραστηριότητες σε συνεργασία με τους άλλους οργανισμούς, τον Eurofound μεταξύ άλλων, διότι... Όλοι εργαζόμαστε προ την ίδια κατεύθυνση από διαφορετική πλευρά όμω. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε και με βάση τα ευρήματά μας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, εξετάζουμε το θέμα της συμμόρφωσής τους. Ε, τι συμμόρφωση βλέπουμε όσον αφορά την ασφαλεία και την υγεία στην εργασία. Και τέλος ε, θα ξεκινήσουμε ε, την έρευνά μας για την έκθεση σε καρκινογενείς παράγοντες. Και Δύο δραστηριότητε που έχουμε προβλέψει για το 2021 είναι αφενό για την κυκλική οικονομία και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Δηλαδή, τι σημαίνει να εργάζεται κανεί στο πλαίσιο αυτή τη οικονομία όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην ε, εργασία. Και επίση μια επισκόπηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Επίση κάτι που ε, πάντα παρακολουθούμε. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Χρειάζεται περισσότερες, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ευαισθητοποίηση για να βελτιώσουμε την κατάσταση σε επίπεδο επιχείρησης. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Δίνω το λόγο στον κύριο Ονεστίνη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τις εργασίες του ETF, του Ευρωπαϊκού Δήματο Επαγγελματικής Εκπαίδευση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την ευκαιρία να σας εξηγήσω τα κυριότερα σημεία όσον αφορά το έργο της υπηρεσίας μας και για να δούμε τώρα αυτά τα σημεία και έχω επίσης φέρει και κάποιες δημοσιεύσεις για να ε, ενημερωθείτε για το έργο μας και όπως γνωρίζετε τα είπαμε πέρσι για μια πρώτη παρουσίαση του οργανισμού με την Επιτροπή είναι ο μόνος οργανισμός και υπηρεσία που λειτουργεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε από αυτές τις πλευράς είμαστε μοναδικοί. Επίσης εορτάζουμε το 19, εορτάσαμε μάλλον την 25η επέτειό μας. Ο, βέβαια θα πρέπει να τροποποιήσουμε ε, το έργο μας, την εντολή μας για να μπορέσουμε να καταφέρουμε καλύτερα αυτά τα οποία μας αντέθηκαν 25 χρόνια πριν, αλλά και για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις ε, αλλαγές, μια που η τελευταία αλλαγή πριν από 10 χρόνια και πάρα πολλοί ε, είπαν ε, τις προτάσεις τους, οι παρατηρητές, Μπάουερ, Σέρκας, επίσης ε, ενεργά συμμετέσχουν και είχαμε προσκεκλημένους από τις χώρες εταίρους όσο μπορούσαν περισσότερους, τους οποίους καλέσαμε, όπως ξέρετε έχουμε 29 χώρες εταίρους από την ε, Μεσόγειο, από Ανατολική Ευρώπη, τόσο από Ανατολική γειτονία μας, από Δυτικά Βαλκάνια, από Αζία και θα για να δούμε τώρα το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμεθα, ε, γιατί πρόκειται για ένα πλαίσιο που σας είναι ε, οικείο. Και Υπάρχουν όλο ένα και περισσότερα κενά σε αυτές τι δεξιότητε και όλο ένα μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των επιχειρήσεων και από την άλλη μεριά ε, του τι παράγει το σύστημα ως ε, δεξιότητες. Σε κάποιες από τις χώρες εταίρου είναι μεγάλο αυτό το χάσμα και ε, εξετάζουμε το ζήτημα του πώ θα αναβαθμιστούν αυτές οι δεξιότητες εκείνες τι χώρε πώς το σύστημα θα εξυγχρονιστεί, γιατί είναι κάτι που σχετίζεται πάρα πολύ με τη βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Οπότε όλη αυτή η κουβέντα είναι σημαντική για να δούμε πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές στην προσπάθειά τους για το μέτωπο αυτό. Κάτι άλλο τώρα, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους εταίρους μας, ε, οι δεξιότητες είναι κάτι που αποκτά μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα. Το είδαμε αυτό στην Ένωση με τον κοινωνικό πυλώνα. Ήταν ένα βασικό επίτευγμα των τελευταίων ετών, κατάρτιση, εκπαίδευση, ανέβηκαν στις προτεραιότητες, αλλά και στους εταίρους μας η υπόθεση αυτή ε, τώρα βρίσκεται στην κορυφή του πολιτικού θεματολόγιου και βλέπουμε και νέα δυναμική όσον αφορά την διεύρυνση. Ε, κάποιοι από τους εταίρους επιταχύνουν τους ρυθμούς τους για να μεταρρυθμίσουν το σύστημα κατάρτισης για να ωφεληθούν από την προσχώρησή τους. Και διαπιστώνουμε στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, όπως έχετε πει και εσείς, ότι θα είναι πολύ βασικό η δεξιότητες και όχι μόνο μέσα στην Ένωση αλλά και στις σχέσεις μας με τους ε, εταίρους γιατί τη βιωσιμότητα προωθεί η Πράσινη Συμφωνία και θέλουμε να υπάρχει βιωσιμότητα και στα σύνορά μας. Οπότε έχουμε αυτές όλες τις ε, συζητήσεις για τα σχετικά προγράμματα. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη βοήθειά μας για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων εκείνων σε εκείνες της χώρας. Αλλά και πέρα από αυτούς και στις χώρες της Αφρικανικής Ένωσης. Να σας πω επιγραμματικά τώρα μερικά αλλά τον Νοέμβριο είχαμε σαντηθεί με κάποιους από εσά και μιλήσαμε για την στρατηγική μας, αν ανταλλάξαμε απόψεις με κάποιους από εσά. Κοιτάξτε, η νέα στρατηγική καλύπτει την κατάρτιση και την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων στις χώρες εκείνες. Αυτό θέλουμε να εξετάσουμε, το πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε τις ικανότητες των χωρών για να προλάβουν και να καλύψουν την αλλαγή στην ζήτηση για τις δεξιότητες στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού συστήματος ευρύτερου και πώς το εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζεται με την αγορά, αλλά τι γίνεται και με το, τι πολιτικές δηλαδή μπορούν να γίνουν. Επίσης δημογραφικές μεταβόλες και μετανάστευση. Επίσης, με τη νέα στρατηγική λαμβάνομαι υπόψη ότι δεν θα πάρουμε νέους πόρους, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο τι προσφέρουμε στους εταίρους. Άρα πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τις χώρες εκείνες που έχουν ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις. Εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δίνουν προτεραιότητα. Και το πλάνο μας είναι να προσφέρουμε εμπειρογνωμοσύνη όπου χρειάζεται. Να δούμε τι θα γίνει τώρα στο μέλλον. Με αυτή την στρατηγική θέλουμε να παγιωθεί ό,τι γνώση έχουμε για να γίνουμε κόμβος γνώσης και αυτά να αξιοποιηθούν και να διαβιβαστούν κατά κάποιο τρόπο να μεταδοθούν στους εταίρους μας. Να συμβουλεύσουμε τις χώρες, να τις βοηθήσουμε και όχι μόνο με προτάσεις αλλά και με το πώς θα υλοποιήσουν τις προτεραιότητες. Άρα χρειάζεται παρακολούθηση, αξιολογία, να λάβουμε υπόψη το ότι στοιχεία υπάρχουν για να προχωρήσουμε σε αυτά τα ε, στοιχεία στρατηγικής. Επίσης πρέπει περισσότερα να κάνουμε συνεργασία και αυτό το οποίο άλλαξε από την αρχή της διαδρομής μας πριν 25 χρόνια είναι ότι τώρα έχουμε πολύ περισσότερους με τους οποίους να συνεργαζόμαστε στα θέματα αρμοδιότητάς μας, διεθνείς φορείς, εθνικοί φορείς, UNESCO, ILO και νέοι εταίροι. Άρα περισσότερη συνεργασία, συνέργεια για να Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα. Δύο λόγια τώρα για φέτος, για το 2020. Είναι μεταβατική χρονιά για να στήσουμε αυτή την καινούργια στρατηγική. Με οριζόντα το τι θα γίνει το 2021 και οπότε έχουμε κάποιες ε, πρωτοβουλίες που τις έχουμε ως σημαίες. Η διαδικασία του Τωρίνου. Έχει σχέση με την εξέταση των ε, εξελίξεων στις ε, χώρες. Το επικεντρωνόμαστε τώρα σε τρεις περιοχές. Ανατολική περιοχή συνεργασίας. Να δούμε επομένως τι γίνεται. Στην ε, Λευκορωσία θα έχουμε μια διάσκεψη για την Ανατολική Γειτονία και και συνάντηση κορυφής αργότερα επίσης ε, χώρες της Μεσογείου και Κεντρική Ασία. Όποιος από εσά ενδιαφέρεται για κάποιο από αυτές τις χώρες είσαστε ευπρόσδεκτοι. Ελάτε να σας πούμε τι πρόγραμμα έχουμε, ας πούμε τις σχετικές ημερομηνίε, οπότε και εσείς να συμμετέχετε σε αυτές όλες τις ζυμώσεις. και θα έχουμε επαφέ με τοπικές αρχές για όλα αυτά τα ζητήματα. Άλλο, γίνονται μελέτες για τις δεξιότητε στο μέλλον. Παραδοσιακή τομή. Να, παράδειγμα. Γεωργία σε Ισραήλ και Μαρόκο, αυτοκινητοβιομηχανία στην Τουρκία, για να δούμε πώς οι ψηφιακές δεξιότητες μπαίνουν σε αυτούς τους παραδοσιακούς τομείς που κυριαρχούν σε αυτές τις χώρες και τι γίνεται όσον αφορά τα αποτελέσματα. Και δούμε τι γίνεται στις χώρες αυτές όσον αφορά τα δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει τόσο καλή οργάνωση των βάσεων δεδομένων όπως τα κράτη-μέλη. Ε, όλα αυτά με το σε σχέση με το τι προοπτικές υπάρχουν για το μέλλον σε αυτό το θέμα, σε αυτές τις χώρες και υπάρχουν και προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κάποιο είδους ε, δίκτυα αριστείας για την κατάρτιση. Οπότε μεταξύ άλλων πέραν των ε, χωρών του έρασμος θέλουμε να καλύψουμε και αυτές τις ε, χώρες εταίρους να μπουν και αυτοί σε αυτή την υπόθεση, να αλλάξει η δυναμική και έτσι. Και έτσι όλες αυτές οι αξίες να προβάλλονται περισσότερο. Και σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Γιονκέριος. Τώρα, έχουμε τώρα την νεότερη των υπηρεσιών και οργανισμών. Την ΕΛΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πράγματι, είναι η πιο πρόσφατη υπηρεσία, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Εργασία, για την Απασχόληση. Άρα δεν μπορώ να μιλήσω για κάποια επέτειο, 25η, οτιδήποτε. Για το 2019 και το 2020 ο βασικός στόχος της αρχής είναι ουσιαστικά να ε, διαρθρωθεί διοικητικά και να στελεχωθεί με προσωπικό η υπηρεσία. Μπορεί να είναι πιο βαρετή η δική μου παρεσίωση σε σχέση με αυτή το προκατόχον, υπό την έννοια ότι ε, εγώ πρέπει να σας μιλήσω για τα logistics. Είχαμε διαδικασίες προσλήψεων για να στελεχωθούμε με επαρκές προσωπικό ώστε να μπορούμε να φέρουμε σε πέρα τα καθήκοντά μας. Υπάρχουν κάποιοι που ήδη εργάζονται για αυτό το τομέα βέβαια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έπρεπε να έχουμε και άλλους. Επίσης είχαμε την καινή θέση για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντού, έκλεισε τα, στα τέλη του προηγούμενου έτους, έχουμε υποψηφίους και θα ακολουθήσουμε τις δέουσες διαδικασίες για τον ορισμό ε, του Διευθυντού που θα αναλάβει καθήκοντα γύρω στο καλοκαίρι του 2020 που σημαίνει, παρόδο ότι μάλλον είναι και η τελευταία φορά που θα δείτε μένα σε αυτή την Επιτροπή. Απ' τη μια αυτό με λυπεί, απ' την άλλη χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό σημαίνει ότι πλέον θα έχει συγκροτηθεί και θα είναι επιχειρησιακή η αρχή για την εργασία. Ένα αυτό. Δεύτερον, είχαμε, κάποιοι ήσασταν παρόντες, στην επίσημη τελετή για την ίδρυση του ΕΛΑ με παρουσία και ευρωβουλευτών και του τότε Προέδρου της Κομισιόν και επίση ε, το Διοικητικό Συμβούλιο ήδη έχει συνεδριάσει δύο φορέ. και ήταν σημαντικό αυτό για τον Οκτώβριο που έγινε και η συγκρότηση του οργανισμού ε, είχαμε και το πρόγραμμα εργασία με το 2018 ε, και πέρυσι το Δεκέμβριο είχαμε μια δεύτερη συνάντηση για το πρόγραμμα εργασίας του 2020 και εκεί εστιάσαμε στις προτεραιότητες του έργου μας για το 2020 με βάση δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διευκόλυνση πρόσβαση ε, σε πληροφορίε για την κινητικότητα, το εργατικό δυναμικό και αποφάσισε το ΔΣ να υπάρξει μια ομάδα εργασία με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να προχωρήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα και έτσι να δοθεί η στρατηγική ενημέρωση που την έχουν ανάγκη οι αρχές και επίσης συντονισμό και υποστήριξη συντονισμένων κοινών επιθεωρήσεων. Θα συνεδριάσει αυτή η ήδη από τον επόμενο μήνα και ελπίζουμε να έχουμε σαφή αποτελέσματα. Ε, βέβαια εδώ πρέπει να έχουμε ένα συμβιβασμό μεταξύ της φιλοδοξίας και του ρεαλισμού γιατί είμαστε στις απαρχές μας, στα σπάργανα είναι αυτή η αρχή. Αλλά τι αποφάσισε η αρχή για την απασχόληση. Να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αδήλωτη Εργασία. Θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενημερωτική εκστρατεία στο πλαίσιο αυτή τη πλατφόρμα. Αποφασίσαμε να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με την πλατφόρμα και σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε κάτι θεωρώ συμβολικό και πολύ σημαντικό ότι δηλαδή θα έχουμε τις πρώτες κοινέ επιθεωρήσεις ε, του χρόνου. Δεν θα είμαστε ακόμα βέβαια σε σταθερή ταχύτητα, αλλά ήδη θα έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά μας και δεν θα μας απασχολούν μόνο τα διοικητικά θέματα, τα υλικοτεχνικά, όσο και αν αυτά είναι σημαντικά, αλλά και επί τόπου θα έχουμε ξεκινήσει το έργο μας για να δείξουμε ότι υπάρχει αυτή η αρχή για την απασχόληση. Το ΔΣ αποφάσισε ε, τις δύο του προτεραιότητες την ενημέρωση αφενός και τις κοινέ ε, επιθεωρήσεις αφετέρου. Δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουμε παραγνωρίσει ή παραμελήσει άλλα σημαντικά πράγματα, τα οποία πράγματι θα μας απασχολήσουν ήδη από φέτος. Να σας αναφέρω δύο εξ αυτών, που είναι και τα πιο σημαντικά να έχουμε την επιχειρηματική συνέχεια για δύο πολύ επιτυχημένα δίκτυα και πλατφόρμες. Το ένα είναι το ΕΟΡΕΣ από την Κομισιόν ε, στην ε, αρχή για την απασχόληση. Ένα δίκτυο που ήδη λειτουργεί και είναι επιτυχημένο θα υπάγεται πλέον στην αρχή για την απασχόληση. Και σίγουρα είναι πολύπλοκη η όλη αυτή η διαδικασία και από Πλευρά ε, μηχανοργάνωση. Θέλουμε να γίνει ομαλά αυτή η μετάβαση. Ένα αυτό. Δεύτερον, νομίζω το είπα και πριν, πλατφόρμα για την αδηλωτή εργασία. Υπάρχει εδώ και δύο χρόνια, όπως ξέρετε, αυτή η πλατφόρμα. Δεν είμαι και βέβαια μερόληπτος γιατί είμαι ο αρμόδιος πρόεδρος αυτής της πλατφόρμας. Νομίζω όμως ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε δεσμεύσει από τα κράτη-μέλη και από τους κοινωνικούς εταίρους. Και όταν γίνει, όπως προβλέπει τρωτικός κανονισμός, η μετάβαση του οργανισμού που πλέον τώρα είναι αυτόνομος και πλέον ε, υπαχθεί στη δική μας την αρχή, ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει την καλή δουλειά που κάνει και βέβαια θα φροντίσουμε γι' αυτό. Ήδη έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και δεν προβλέπω να αντιμετωπίζουμε ιδίω για τη δεύτερη μετάβαση και για την πρώτη κάποια δυσκολία. Με ενθαρρύνει άλλωστε ιδιαίτερα και το γεγονό ότι και η πλατφόρμα και η αρχή ήδη συνεργάζονται. Όπω είπα και στην αρχή. Έχουμε και προκλήσει βέβαια να αντιμετωπίσουμε για το χρόνο και τα επόμενα έτη. Τώρα, Ίσως η φιλοξενία των εθνικών συνδέσμων θα είναι ένα πρόβλημα από διοικητική υλικοτεχνικής πλευράς. Αυτοί οι σύνδεσμοι έχουν ένα σημαντικό ρόλο για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας μας και ελπίζουμε στο πρώτο εξάμεινο του έτους να έχουμε ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και βασιζόμαστε σε αυτούς. Τα κράτη-μέλη πρέπει όμως να ορίσουν τα σωστά άτομα, τους πιο ικανούς και κατάλληλους για αυτή τη θέση και φαντάζομαι ότι θα γίνει. Με το ΔΣ έχουμε συμφωνήσει σε ό,τι αφορά την περιγραφή εργασίας και το προφίλ των ατόμων αυτών. Θέλουμε βέβαια αυτοί οι άνθρωποι να διατηρήσουν με ισχυρού δεσμού με την εθνική δίκαιση, αλλά να εργάζονται επίση και στο πλαίσιο το ενωσιακό. Στο πλαίσιο τη αρχή για την απασχόληση. Έχουμε λοιπόν αφενός τα θέματα τελικοτεχνικά, υποδομών, επιμελητίας. Οι μη πολιτικοί γνωρίζουμε ότι αν δεν λειτουργούν αυτά έχουμε πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ισορροπήσουμε πάνω σε ένα λεπτό σκηνή, γιατί θα είμαστε πλέον επιχειρησιακοί το 2020 και πρέπει να ρυθμίσουμε και άλλα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει λάβει προτάσεις και θα λάβει και άλλες προτάσεις, κυρίως ό,τι αφορά αυτές τις ε, κοινέ επιθεωρήσεις που θα οργανωθούν. Να σας ε, πω ανεκδοτικά και κάτι που συνέβη σε αυτό το ΔΣ. Είχαμε προτείνει να υπάρξει τουλάχιστον μια κοινή ε, επιθεώρηση. Εμείς, αλλά το ΔΣ είπε όχι μόνο μία και άλλες να κάνετε. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Θα δώσω τώρα το λόγο, καταρχάς στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ε, ίσως να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα σε ένα γύρο. Πρώτα από το ΕΛΚ η κυρία Φρανσόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις ε, ε, παρουσιάσεις, τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για, τις, για τη δουλειά που κάνουν οι διάφοροι οργανισμοί. Είναι πολύ χρήσιμες για τις εργασίες μας οι στατιστικές και προσβλέπουμε στην συνέχιση της καλής συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή ΕΜΠΛ και τους οργανισμούς αυτούς, καθώς και με την Νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Κυρία Πρόεδρε, ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να επισκεφτούμε τις, ε, τους ε, οργανισμούς κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας, τους νέους οργανισμούς. Και δύο ερωτήσεις. Πώς μπορούμε καλύτερα να ενσωματώσουμε τις ε, συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στις αποφάσεις μας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι... Θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε την αίσθηση ότι αυξάνεται ο φόρτος εργασίας των οργανισμών σας και ε, είναι επαρκής ο προϋπολογισμός. Μπορώ να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση αμέσως, διότι συνήθως επισκεφτόμαστε κάθε χρόνο έναν οργανισμό. Και ρωτάμε ποια μέλη της Επιτροπής μας θέλουν να συμμετάσχουν. Μαρία Φίντα από το S&D. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, σύντομες αλλά πολύ σημαντικές ε, παρουσιάσεις σας. Ε, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά για την Ευρώπη. Θα συνεχίσω στα Δανέζικα, λέει ο Μιλήτρια. Κύριε Σίπελ, είναι πολύ σημαντικό όλοι στην Ευρώπη να λαμβάνουν κάποια μορφή ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό όλοι να καταλάβουν πώς μπορεί να αλλάξει ο χώρος εργασίας ε, για να ευημερούν οι εργαζόμενοι. Πώς ε, βλέπετε εσείς το στόχο ε, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια όλοι στην Ευρώπη να έχουν μετακπαίδευση. Κύριε Μενέντες Βαλτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, πολύ πλήρη παρουσίαση της Eurofound. εγώ είμαι χρήστης, χρησιμοποιώ πολύ συχνά την ιστοσελίδα σας, περιέχει πάρα πολλά στοιχεία. Αναφερθήκατε στην ε, διαφάνεια όσον αφορά τις αμοιβέ. Ε, ε, ξέρω ότι άντρες και γυναίκες δεν λαμβάνουν την ίδια αμοιβή στην Ευρώπη. Η διαφάνεια θα βοηθήσει και ε, κυρία Λάτσεκ, ήμουνα, κυρία Σετλάτσεκ, ήμουνα ε, στην Κοπενχάγη στην παρουσίασή σας ε, για τις ε, επικίνδυνε ουσίες. Ο τρόπος δηλαδή που ενσωματώσατε παραδείγματα από την πραγματική ζωή, από τους χώρους εργασίας στις παρουσιάσεις σας, ενέπνευσαν όλους και όλοι επέστρεψαν στους χώρους εργασίας τους και αλλάξαν τα πράγματα. Ελπίζω να κάνετε το ίδιο όσον αφορά τι μειοσκελετικέ διαταραχέ. Το να δούμε δηλαδή ότι υπάρχουν επιχειρήσει που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, αυτά αυτό καν, αλλάζει την οτροπία αυτών που ακούνε ε, τα στοιχεία αυτά. Ο ε, κύριος Σίπελα αναφέρθηκε στις αλλαγές στον χώρο εργασίας. Ε, ε, αν δεν είναι κανείς προετοιμασμένος, ε, αν δεν είναι κανείς ε, προετοιμασμένος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ψυχοσωματικά προβλήματα, σε πολύ υψηλά επίπεδα στρες. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το θέμα αυτό ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Μπρινέ από το Ρενιού. Μπορώ να της δώσω το λόγο ή να δώσουμε το λόγο σε κάποιον άλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παραχωρώ τη θέση μου στην Βερονίκη Λενόρ που έχει ένα συγκεκριμένο ερώτημα στον τομέα της υγείας. Τρίλε Λενουάρ, να σας τα πω στα γαλλικά λέει η κυρία Λενουάρ. Οι ερωτήσει μου αφαιρούν την κυρία Σέντλατζεκ όσον αφορά την υγεία στον χώρο εργασίας. είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις καρκινογόνες ουσίες. Οι πολύτιμοι έχουμε. έχουν. 120.000 είναι οι καρκίνοι που διαγνώσκονται κάθε χρόνο. Και ε, αυτό αντιστοιχεί σε 80.000 θανάτους. Και η αγωγή έχει προχωρήσει η ιατρική, αλλά πάρα πολύ ε, έχουν προβλήματα μετά να επανταχθούν στο εργασία από του ασθενήσαντε. Μήπως μπορούμε να δούμε διάφορα στοιχεία για την εργασία και να δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αυτά θα μπορούσαν να προσθεθούν στον χάρτη πορείας που έχετε για τις καρκινές ουσίες. Επίσης, να σας πω για μια ανησυχία μας όσον αφορά αυτές τις ε, καρκινές ουσίες που δεν έχουν σχέση με το περιβάλλον γιατί μεταξύ αυτών ξέρετε ότι έγινε μία μελέτη και καταλήξανε ότι κινούν περισσότερο γυναίκε με καρκίνο του στήθους να δουλεύουν τη νύχτα. Και επίση χρειάζεται τελικά να υπάρχει μια εκστρατεία για να υπάρχει ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που οδηγούν σε καρκίνο αλλά χωρίς να έχουν σχέση με ουσίες ε, σχετικές με το περιβάλλον. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Από τους πρασίνους. Όχι. ID. Κύριε Κόκκιν, θα λάβετε το λόγο για το ECR. Δυστυχώ, ε, μόλις ε, κατέφτασα διότι είχα μια διάσκεψη πριν ε, και γι' αυτό δεν έχω μπει καλά στο θέμα. E. Ούτε βλέπω κάποιον από την ΚΟΕ. E. Να ακολουθήσω τότε τον κατάλογο όσων ζητούν το λόγο και κατόπιν θα λάβετε κι εσείς ε, το λόγο. Πρώτα λοιπόν τους ευρωβουλευτές, μετά τους εμπειρογνώμονες και μετά στους διευθυντές. Θα δώσουμε πάλι τον λόγο. Γιώχαν Τάνιελσεν πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους ε, για τις παρουσιάσεις ε, των προγραμμάτων εργασίας των οργανισμών. Δύο ερωτήσεις έχω σχετικά με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Καταρχάς, επικροτώ το ότι θα δώσετε προτεραιότητα στις κοινέ επιθεωρήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση θα είχε να κάνει με, την, με τις φιλοδοξίες στα πιλωτικά προγράμματα για να γίνει τουλάχιστον μία πιλωτική επιθεώρηση, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είσαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι και σας ε, καλώ να το κάνετε ακόμη περισσότερο. Θα ε, ε, το επικροτήσω ιδιαίτερα αν έχετε πάνω από μία τέτοια επιθεώρηση. Νομίζω ότι μία επιθεώρηση για ένα χρόνο είναι αρκετά περιορισμένη φιλοδοξία. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω τι συνέργειες υπάρχουν με υπάρχοντες φορείς και σε εθνικό επίπεδο για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να αποφευθεί η αλληλεπικάλυψη στις δομές. Ε, με μια δεύτερη ερώτηση έχω ε, για άλλο τμήμα της ε, δουλειάς του οργανισμού. Στο άρθρο 8 του κανονισμού λέει ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να εφιστούν την προσοχή της ε, αρχή ε, σε διάφορες υποθέσεις. Και ήδη κατά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ε, είχαν υποβληθεί διάφορες υποθέσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μέσω της ΕΤΥΚ. Φέτος λοιπόν, ε, τι συγκεκριμένα μέτρα ε, σκοπεύετε να λάβετε όσον αφορά τις εκκρεμούσε αυτές τις υποθέσεις, ε, καθώς και τις νέες υποθέσεις που θα εμφανιστούν. Ευχαριστώ, Ντουινά Φερνάντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να σας τα πω καλύτερα στα ισπανικά πρώτα-πρώτα. Εννοείται ότι ευχαριστούμε τους εκπροσώπους των υπηρεσιών και οργανισμών και αυτό που θέλω να ρωτήσω αφορά τον κύριο Μενέντεθ Βάλτες αλλά και την κυρία Σεντάλσκι για τα θέματα της υγείας. Όντως, μπράβο για όλες αυτές τις ε, μελέτες που έχετε οργανώσει και αναλάβει όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας ε, για να βοηθήσετε το θέμα της υγείας και εργασίας. Αλλά υπάρχει εδώ ε, ένα κενό, το ζήτημα της πνευματικής υγείας στο χώρο εργασίας και σας τονίζω, γιατί τα έχουμε πει ναι, και σε άλλες συναντήσεις μας ε, αφορά τις κοινέ διαταραχές ε, σε σχέση με κατάθλιψη ή με προβλήματα προσαρμογής. Αυτές οι διαταραχές έχουν σχέση με συγκεκριμένο περιβάλλον, με συγκεκριμένη ε, συγκυρία στην δουλειά. Οπότε αυτές τους διαταραχές σχετίζονται γενικότερα με το κατά πόσο κανείς επιμελείται την υγεία. Ε, και αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη είναι ευρωπαϊκή στρατηγική για την διανοητική υγεία. Γιατί υπάρχουν σχιζοφρένειες και άλλες σοβαρές διαταραχές και εγώ εργάζομαι σε μια επιτροπή που το, το θέμα μας είναι οι κοινέ διαταραχές. Τι πρόληψη μπορεί να υπάρχει ε, ε, επομένως πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να εντοπιστούν οι εργασιακές συνθήκες που βοηθούν στο να υπάρχει καλύτερη διανοητική υγεία απλώ οργανωμένων. Και είναι αλήθεια ότι έχετε εκπονήσει πολλές μελέτες, αλλά χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και περισσότερη πίεση, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο που μας πρόσκειται το θέμα, να δώσουμε συστάσεις σε όλα τα κράτη για τις εργασιακές συνθήκες που βοηθούν στο θέμα της διανοητικής υγείας. Ε, ο πλευράς ψυχοκοινωνικής που είναι βασικό και όπως και εσείς επισημάνατε υπάρχει το θέμα της ψηφιοποίησης που επίσης σχετίζεται και επηρεάζει ε, στο επίπεδο αυτό η υπερσυνδεσιμότητα και άρα χρειάζεται να υπάρξει σχετική νομοθεσία και προσπαθούμε εμείς από την Επιτροπή μας όσον αφορά την αποσύνδεση ε, γιατί έτσι προλαμβαίνουμε τέ, τέτοιες διαταραχές, τέτοιες ε, αρρώστιες και αυτό θα οδηγήσει σε, λιγότερο απουσιασμό ακόμα και σε λιγότερες αυτοκτονίες. Άρα σας ευχαριστώ για όσα κάνετε αλλά συνεχίζω να σας ζητώ να πασχίζετε και να βοηθήσετε το έργο του Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο γιατί άρα χρειάζονται καινούργια μοντέλα για τις συνθήκες εργασίας που να βοηθάνε όχι μόνο τη σωματική αλλά και την διανοητική ψυχική υγεία. ευχαριστούμε. Πέτερ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχω κάτι κοινό με τον κύριο Κορέλ και τον κύριο Μενέντες Βάλτερ. Ότι είναι και η δική μου τελευταία φορά εδώ στην Επιτροπή. Θέλω να σας ευχαριστώ και λοιπόν για το εξαιρετικό σας έργο και να σας ευχηθώ καλή τύχη από εδώ και πέρα. Επίσης τον κύριο Νεστίνη. Γειτονική χώρα θα είμαστε. Θα έρθετε στη Βρετανία. Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω. Από την Ιρλανδία. Ε, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε 75 εκατομμύρια Ευρωπαίου στο εργατικό δυναμικό, οι οποίοι δεν έχουν υψηλέ δεξιότητε, ένα στου τρει δηλαδή, και μιλάμε πάρα πολύ για του νέου. Όμω, εγώ είμαι ε, μεγαλύτερος. Με ενδιαφέρουν και αλλαγέ δημογραφικές για τον πιο γύρω πληθυσμό. Τι θα γίνει με την παιδεία, την εργασία και την απασχόληση και τις διάφορες ισορροπίες και συσχετισμούς. Πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και στρέφομαι εδώ στον κύριο Ζίμπελ. Τι γίνεται από αυτού. Ε, τι δουλειά κάνει σε ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Έχετε κάποια συμμετοχή στο πρόγραμμα φιλικών πόλεων τη... της Κομισιόν. Θα ήθελε και η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς βέβαια να συγχαρώ ε, τους πέντε διευθυντές. Ο κύριος Ζιμπελ πολύ σωστά είπε ότι είναι πρόκληση. Γιατί υπήρχαν τέσσερις οργανισμοί, τώρα υπάρχει ο πέμπτη, ο αυτή αδελφή εντός αγωγικών ε, νέα υπηρεσία Άλλοι έχετε εντολή ε, εδώ και 25 χρόνια, κάποιον έχει επικαιροποιηθεί. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να επανακαθοριστεί η ε, διαχωρισμός εργασίας για να μην υπάρχουν λυπικαλύψεις, να ε, επανεξεταστεί η εντολή αυτών των πέντε πλέον οργανισμών. Ένα ερώτημα αυτό και δεύτερο. Θα με ενδιαφέρει να είναι πολύ έτσι, ισχυρή η δημόσια υπηρεσία στην Ένωση. Αλλά ξέρω ότι έχετε σφιχτού προπολογισμού και δεν μπορούσατε να απασχολήσετε περισσότερο προσωπικό, θα προσλάβετε νέα άτομα. Και υπήρχε τάση σε πολλού οργανισμού να προσλαμβάνουν προσωρινώ απασχολούμενου συμβασιούχου ή να αναθέτουν σε εξωτερικού συνεργάτε πολλέ εργασίε. Είναι μια τάση τη εποχή και θα ήθελα να ξέρω στι υπηρεσίε σα ποιοι είναι αυτοί που έχουν, πόσοι είναι αυτοί που έχουν καλές μόνιμες συμβάσεις και δηλαδή, σε τι αναλογία σε σχέση με τους συμβασίους και λοιπούς. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει. Η πρώτη αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Απασχόληση. Έχουμε πολλές προσδοκίες και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον η αρχή αυτή έχει ήδη επιληφθεί κάποιων θεμάτων, αν έχει πάρει κάποια αλληλογραφία ήδη και αν ναι, γιατί θέματα. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά ιδίως ε, το ΣΕΝΤΕΦΟΠ για τα προσόντα, για τα μελλοντικά προσόντα και δεξιότητες της χώρες Μεσογείου. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τι κάνετε ιδίω για τι επιχειρήσεις επαγγελματικού τομεί για να ε, ξέρουμε λίγο πολύ τι, ποιες θα είναι οι μελλοντικέ ανάγκες σε δεξιότητες και προσόντα. Ευχαριστώ. Τέλος, λέει πρόεδρος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μίλλερ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες που λάβαμε. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τις παρουσιάσεις σας. Ε, ιδιαίτερα με ενδιέφεραν οι προσπάθειες που αναφέρατε για προσαρμογή των ε, για προσαρμογή στις ανάγκες ε, της αγοράς εργασίας ε, και αυτό δεν είναι κάτι νέο, είναι κάτι που το ακούμε ε, εδώ και κάποια χρόνια. Ο συντονισμός δηλαδή του συστήματος κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας δεν είναι κάτι νέο. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε πώς έχει εξελιχθεί το θέμα αυτό σε βάθος χρόνου. Βελτιώνεται ο συντονισμός διότι από τη μία αναλύουμε την αγορά εργασίας, διαπιστώνουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε δεξιότητες, αλλά μπορεί να υπάρχει κενό ανάμεσα σε αυτά που κάνετε εσείς και τις ανάγκες της αγοράς. Η δουλειά σας είναι αποκλειστικά θεωρητική Σκοπός είναι απλά να γίνονται έρευνες ε, ή προσαρμόζεστε στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νόμιζα ότι είχαμε κλείσει με τους ευρωβουλευτές. Ε, ε, Δίνω το λόγο στην κυρία Ρέγνερ και μετά ε, θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Ε, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που με επιτρέπετε και εμένα να θέσω μια ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με την ισότητα των δύο φύλων ε, και απευθύνομαι σε όλους τους διευθυντές. Πώς εφαρμόζεται την ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων στον δικό σας οργανισμό. Δεύτερον, σε τι βαθμό Έχετε καλή συνεργασία και με την ΑΕΝΚΕ, τον, ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για ε, την ισότητα των δύο Όσον αφορά το Ίδρυμα του Δουβλίνου, καταλαβαίνω ότι πολλά συνδυάζονται. Ε, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, οποιασδήποτε συνέργειες πιθανόν να υπάρχουν και επίσης γενικά βλέπω Ε, το θέμα των ε, εργαζόμενων ε, γυναικών. Ανακύπτει λοιπόν το θέμα του, της διαφοράς στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών και ιδιαίτερα από τον οργανισμό του Δουβλίνου θα ήθελα να ακούσω σε τι βαθμό Ε, ετοιμάζεστε για τις εργασίες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και όσον αφορά τον ελάχιστο μισθό, πολύ συχνά οι γυναίκες κατέχουν τις θέσεις της, με τη χαμηλότερη αμοιβή. τι κάνουν λοιπόν οι οργανισμοί σας. Ζητώ συγγνώμη που τώρα στο τέλος έθεσα τις ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ Εβελίν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο Ε, στον πρώην συνάδελφο Μπέκερ που είναι εμπειρογνώμων μας στην ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Σίπελ για την επισκόπηση ε, της παρούσας φάσης εργασίας μας. Γνωρίζουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και από τις δημογραφικές εξελίξεις. Ε, είναι λοιπόν σημαντικές οι πτυχές αυτές. και οι ε, πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και η διαβίου μάθηση είναι σημαντικά θέματα λαμβάνοντας υπόψη και την ε, ε, έλλειψη σε εξειδικευμένους εργαζομένους που αντιμετωπίζουμε. Η τεχνογνωσία του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντική ώστε να εντοπίσουμε τους τομείς όπου θα πρέπει ε, να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες. Στις ε, στρατηγικές παρουσιάσεις ε, το θέμα είναι πώς μπορούμε να ασκήσουμε πίεση ή να το πω πιο γενικά πώς μπορούμε να κοινοτοποιήσουμε τις εθνικές κυβερνήσεις, τους εθνικούς οργανισμούς, αρμόδιους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους που όπως γνωρίζουμε παίζουν πολύ επικοδομητικό ρόλο. Πώς μπορούμε λοιπόν να τους κινητοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο να καταβάλουν προσπάθειες. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών ε, για ε, ένα νέο σύγχρονο όραμα του χώρου εργασίας ε, είναι επίσης κάτι σημαντικό. Ε, η διαβίου μάθηση είναι πολύ σημαντική. Και υπαρξιακό ερώτημα σχεδόν για την Ευρώπη είναι και σας περιγράφω πώς βλέπω εγώ τη δική μου δουλειά ως εμπειρογνώμων στο μέλλον. Το υπαρξιακό λοιπόν είναι ακριβώς οι δεξιότητες, η εξειδίκευση των εργαζομένων. Ε, θα πρέπει να βρισκόμαστε στην κορυφή στο θέμα αυτό. Καλό λοιπόν όλους τους συναδέρφους ε, της Επιτροπής ΕΜΠΛ να στηρίξουν ε, τέτοιες εργασίες. Ένα σύνθημα που άκουσα πρόσφατα ήταν το «Making VET fit for the future». Σα Σας ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λόπες Φοντενέιρα που είναι πυρογνώμων μας στον Eurofound. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς όπως είπε ο κύριος Μενέντες Βάλτες, ο στόχος της υπηρεσίας είναι το να βοηθά Ευρωπαϊκό Οργανισμό, Εθνικό Οργανισμό με κάποια δεδομένα, με κάποια συμπεράσματα που δεν μπορούν τη λήψη αποφάσεων. Όσα μα είπε ο Μενέντε ήταν πάρα πολύ σαφή και διαπιστώσαμε το σπουδαίο έργο των υπηρεσιών αυτών τα τελευταία χρόνια. Και εγώ είμαι παλαιά βουλευτή και γνωρίζω τι δυσκολίε ε, τη ε, νομοθεσία για τη βελτίωση των ε, βιωτικών συνθήκων και εργασιακών συνθήκων ε, και σε επίπεδο προσωπικό και εργασιακό. Ε, Επομένω, έχουμε ε, αντικειμενικές πληροφορίες βάσει δεδομένων, τι αναλύσεις συγκεκριμένων ομάδων, συνέπειες επιπτώσεις πολιτικών, οπότε έτσι τα πράγματα γίνονται ευκολότερα. Αυτά που μας δίνει το Eurofund είναι ό,τι χρειάζεται ακριβώς όπως ε, εξηγήθηκε σε σχέση με τον ελάχιστο μισθό που είναι θέμα της καυτής επικαιρότητα και είναι θέμα τόσο επίμαχο. Επομένως θα πρέπει όλα αυτά προσεκτικά να τα αναλύσουμε ακριβώς και στα πλαίσια ε, του άλλου θέματος που έχουμε για τη σύνθεση των οικοκυριών και τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε μια γενικευμένη βελτίωση στην αγορά εργασία της ε, Ένωσης. Παραμένουν πάντως οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ χωρών, περιφερειών και υπάρχει στον ορίζοντα απειλή διαταραχής της οικονομικής ε, συγκυρίας. Οπότε έχουμε και σημαντικούς δημογραφικούς στόχους, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την κλιματική αλλαγή. Σίγουρα πάντως ε, χρειάζονται κάποια δεδομένα ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας για όλους αυτούς τους ε, στόχους και θα πρέπει βέβαια να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η έρευνα που γίνεται και αυτό απαιτεί πρικοδότηση. Αλλιώς θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες όπως είπαν διάφοροι συνάδελφοι όσον αφορά την υπεργολαβία του έργου των υπηρεσιών, που είναι θέμα οικονομικό. Άρα, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστήριξει τις υπηρεσίες αυτές, ούτως ώστε να έχουν τον προπολισμό που χρειάζεται. Επίσης, ολοκληρώνω επενθυμίζοντας ότι καταστροφή απασχόλησης σημαίνει δημιουργία απασχόλησης, θέσεων εργασίας δηλαδή, να υπάρχει ποιότητα, ανταγωνιστικότητα, ε, βελτίωση των επιδόσεων όσον το κόστος αλλά και προστασία των εργαζομένων. Επίσης, μπράβο στον κύριο Μενέντες για το έργο του τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μίκητσο Είστε ο μας της όσα. Ε, Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το προσωπικό της ε, υπηρεσίας γιατί με καλοδέχτηκαν ε, τέλος της προηγούμενης εβδομάδας από πλευράς του, Διευθυντικού Συμβουλίου. Ε, αυτό είναι καλή αρχή. Και επίσης χαιρετίζω τις προτεραιότητες που η υπηρεσία όρισε για του χρόνου, ψηφιοποίηση, ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία, Ήδη η δόκτωρ Σέντλουτσεκ μας τα είπε για το ψυχοκοινωνικό κίνδυνο που αναφέρθηκε από κάποια βουλευτή και είναι σημαντική προτεραιότητα για όλους μας να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε το θέμα των προτεραιοτήτων όπως τα είπαν οι βουλευτές και να τις εντάξουμε στο πρόγραμμα εργασίας της υπηρεσίας. Το μπορούσα να πω ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο τα θέματα που έχουν σχέση με τον καρκίνο. Όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Δηλαδή, ποια στοιχεία στη δουλειά σχετίζονται με την ασθένεια. Πρόκειται για προτεραιότητα. Το έταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προτεραιότητα και είναι πολύ σημαντικό το θέμα και για την Επιτροπή σας. Θα πρέπει και για τη δική μας δουλειά επίσης να είναι προτεραιότητα. Τώρα, για τον χρόνο έχουμε τρεις προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. είναι η αρχή της εργασίας μας παρά όλα αυτά. Επισήμανα τις εξής προκλήσεις. Πρώτον, κάτι το οποίο ήδη έχει ληφθεί υπόψη από την υπηρεσία να προσπαθήσουμε να καλύψουμε και να έχουμε επαφή με τις ε, μικρές επιχειρήσεις και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Να συνεργαστούμε με τους εθνικούς κόμβους που ασχολούνται με το ζήτημα, για την βοήθεια αυτών των επιχειρήσεων, γιατί είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Οπότε συνεργαζόμαστε επομένω με αυτά τα γραφεία στα κρατημέλη και αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει τα κρατημέλη Θα πρέπει αυτή η συνεργασία να είναι απαλλαγμένη από γραφειοκρατία, να λειτουργεί πιο εύρεθμα. Αυτό μπορεί να το φροντίσει και η όσα. Πάντως για το άμεσο μέλλον το πιο σημαντικό είναι να επεξεργαστούμε την ευρωπαϊκή στρατηγική για ασφάλεια και υγεία στη δουλειά. Εμείς θα συμβάλλουμε πολύ. Και η Επιτροπή επίσης θα βοηθήσει και θα συμβάλλει ε, Τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιήσαμε βασίζονται σε ερωτηματολόγια, σε έρευνα 50.000 ε, συμμετεχόντων. Αυτά. Έχω δύο από το ETF Σέρκας, καταρχάς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους και από την Επιτροπή και αυτούς που ε, είναι εδώ και από τους οργανισμούς. Ήμουν και εγώ ευρωβουλευτής και τίμησα το έργο όλων. Τον κύριο Μενέντες Φαλτές που τον αποχαιρετούμε σήμερα ε, πρέπει να πω ότι βλέπω, παρότι είμαι πλέον εκτός κοινοβουλίου, ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ είμαι στο Τωρίνο, στο ETF. Θέλω να πω ότι όσο ήμουν ε, στις συνεδριάσεις ως παρατηρητής στο Τωρίνο και αλλού, εκτίμησα την πολύ καλή δουλειά που κάνουν με πολύ λίγα κονδύλια 29 χώρες. Και δεν ξέρω πραγματικά πώς να το πιστέψω μερικές φορές. Γιατί πραγματικά βοηθούν πολύ. Όταν θέλουμε να αυξήσουμε την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου σε χώρες που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Το Τωρίνο λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ως οργανισμός. Θέλω να πω τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ φορέ οι φιλοδοξίε μα ξεπερνούν τα μέσα που έχουν στη θέση μα και αυτό ε, δημιουργεί απογοητεύσει που πώ μπορούμε να τι υπερκεράσουμε αν αυξήσουμε τη δουλειά μα και την ποιότητα τη δουλειά. Είπε ο Διευθυντή ότι έχει νέα φιλοδοξίε και νέα στρατηγική. Αν οι πόροι δεν αυξηθούν όμως, δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ εύκολο και πρέπει και εσείς οι βουλευτές Επιτρόπης Απασχόλησης να κάνετε ό,τι μπορέσετε. Και στο πλαίσιο των ετήσιων προπλησμών και των δημοσιονομικών προοπτικών. Γιατί αν δεν έχουμε μαζί με τις φιλοδοξίες επαρκή χρηματοδότηση θα προκύψει εκ νέου απογοήτευση. Και επαναλαμβάνω, 29 χώρες ε, βοηθά το ETF, το το Ίδρυμα για την Εκπαίδευση. Υπάρχει μια νέα στρατηγική μετά τα 25 αυτά χρόνια. Ε, μια νέα φάση ξεκινά. Και πρέπει να υπάρξουν περισσότερες συνέργειες ε, να συνεργαστείτε με πολλούς άλλους φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαβιούμάθηση και της εκπαίδευσης. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά αυτές οι ενώσεις ή άλλοι φορείς ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια των 29 ετών. Τι θα γίνει με τους Βρετάνους, θα τους αφήσουμε μόνος τους με αυτή τη μεγάλη τεράστια τρύπα που ανοίγει τώρα. Και να πω επίσης ολοκληρώνοντας ότι πραγματικά έμαθα πάρα πολλά από τις συναντήσεις μου με συναντήσεις μας στο Τωρίνο. Εκτιμώ όλος ε, την αφοσίωση και τις ικανότητες ε, του προσωπικού σας και θέλω εξ ονόματος μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για όλους σας. Πραγματικά είναι ε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των νοσιακών θεσμών στις χώρες μέλη αυτοί οι οργανισμοί. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να με ακρηγορήσω, θα τα πω στα σλοβακικά. Πριν περάσω σε κάποιες παρατηρήσεις, ερωτήσεις, θα ήθελα να σας πω το εξής. Στην Επιτροπή μας είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους οργανισμούς που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Και αυτό ισχύει και για τους συναδέλφους που είναι εδώ. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε, οι ευρωβουλευτές μπορούν να είναι περήφανοι για τους ε, οργανισμούς. Εκτός από τον ΕΛΑ, ε, την αρχή για την απασχόληση, είχαμε επαφές με όλους τους άλλους ε, οργανισμούς. Ε, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία για τις κοινέ αυτές επιθεωρήσεις πριν από 10 χρόνια θα ήταν κάτι που ούτε θα μπορούσαμε να το φανταστούμε. Και σήμερα είναι πραγματικότητα που σημαίνει ότι σιγά σιγά έχουμε πλέον σημειώσει επιτυχίες. Αν μου επιτρέπετε τέσσερις ερωτήσεις για το ETF που πολλές φορές είναι στο περιθώριο. Δεν το προσέχουμε τόσο πολύ στην Επιτροπή μας. Δεν είναι δηλαδή η ε, προβολή στραμμένη πάνω του. Παρόλα αυτά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Υπάρχει μια επικέντρωση σε τρίτα κράτη. Οπότε δεν ξέρω αν και η Επιτροπή για την Ανάπτυξη, την Περιφερειακή Ανάπτυξη θα έπρεπε να επιληφθεί Γιατί έτσι πιστεύω ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι πιο πολύ το πεδίο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη, κατά δεύτερον. Εδώ πραγματικά έχουμε σημαντική εμπειρία. Έχετε 25 ετή εμπειρία και σε αυτό το πλαίσιο Έχετε πολύ ασχοληθεί με την επαγγελματική εκπαίδευση. Εγώ θέλω να μιλήσω από προσωπική εμπειρία, προσωπική πείρα. Στα κράτη-μέλη ε, δεν αξιοποιούνται παρκώ οι εμπειρίε σα όπω θα έπρεπε και αυτό είναι κρίμα. Τρίτη παρατήρηση ερώτηση. Είναι ένα, ή θέλουμε να γίνει ένα παγκόσμιο πρωταγωνιστή αυτό το ETF. όμως συμμετέχετε στην χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής και έχετε συνεργαστεί με πολλές τρίτες χώρες. Τώρα συνεργάζεστε ή τέλο πάντων ε, ασχολείστε με 29 κράτη και θα έχετε πλέον ε, συμμετοχή και στις εργασίες ε, της Παναφρικανικής Ένωσης. Δεν ξέρω αν είναι θετικό ε, το να θέλουμε να δώσουμε ένα δις για την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά το ETF να έχει όλο και μικρότερο προπολογισμό κάθε χρόνο, που ασχολείται και με αυτή την πτυχή, άρα είναι κρίμα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας και τις δραστηριότητες που προβλέπονται κάθε δύο μέρες η Κομισιόν θέτει νέες απαιτήσει ε, και πρόκειται για σίγουρα άκρος ποιοτικό έργο. Υπάρχει και τρομερό φόρτος εργασίας ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό ε, να αντιμετωπιστεί από πλευράς Κομισιόν. Δεν συνδυάζεται όλο και περισσότερα καθήκοντα, όλο και λιγότερα χρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τέλος, Αρκ ε, πυρογνώμων του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρόσφατα συζητήσαμε τις διαπραγματεύσεις για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Και τώρα ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε μέσα Οκτωβρίου και μέσα σε τρεις μήνες, όπως ήδη μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε δύο συναντήσεις όπου συμμετείχα ως προσκεκλημένος, διότι δεν είχε γίνει επίσημος διορισμός ακόμη. Τρει μήνε είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να αξιολογήσει κανεί τα όσα συμβαίνουν, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο. όσον αφορά αυτό το πρώτο διάστημα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να καταργήσει πολλές ε, τυπικές διαδικασίες. Ε, θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο με πολλές διαδικασίες κλπ. Εγώ τα έχω καταγράψει αυτά ε, ε, σε δύο σελίδες που σας έχω υποβάλει. Δεν χρειάζεται να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Πάντως, σε πολύ σύντομα θα έχουμε ένα επόμενο βήμα. Δύο ομάδες εργασίας θα ξεκινήσουν τις εργασίες τους ε, την επόμενη εβδομάδα και κατόπιν βήμα-βήμα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, κάνοντας ε, πρωτοποριακή δουλειά. Ε, Αρκετές προκλήσεις αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, η ομαλή μετάβαση, η συμπερίληψη όλων των θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, πολλές επιθυμίες που εκφράσαμε ε, εδώ στο Κοινοβούλιο καθ' όλη τη διάρκεια των ετών ε, για να ε, αποφύγουμε να αντιμετωπίζουμε τα θέματα σε στεγανά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή το να μην ξεκινήσουμε από το μηδέν, διότι υπάρχουν αρκετέ πρωτοβουλίε εντό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Υπάρχει και αρκετή ε, διακρατική συνεργασία ανάμεσα σε ε, επιθεωρητές εργασίας. Αξίζει τον κόπο να τα κοιτάξουμε αυτά και να τα ενσωματώσουμε στι εργασίε τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνο αν υπάρχουν υπερβολικά πολλοί στόχοι, να μην επιτυγχάνεται κανείς από αυτούς. Ε, είναι σοβαρός αυτός ο κίνδυνος. Η βασική πρόκληση όμως είναι πώς να διευκολύνουμε και να διευκολύνουμε τις εργασίες όλων των εθνικών παραγόντων που ε, έχουν να κάνουν ε, με την κινητικότητα και τα σχετικά δικαιώματα. Οι παράγοντες αυτοί είναι πολύ και διάφοροι. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Γιόν. θα είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας ε, καλός μηχανισμός ε, συναγερμού, ε, κοινοποιήσεων, Αυτό δεν ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό. Πρόεδρε, αυτά έχω να σας πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις ακούσαμε. Σας δίνω το λόγο με την ίδια σειρά που σας τον έδωσα αρχικά και ελπίζω να μπορέσετε ε, να απαντήσετε. Ωραία. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να ε, απαντήσω σε αυτές που αφορούν ε, τον ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Θα ξεκινήσω από την κυρία Φίντ. τι πληροφορίες παρέχουμε στους πολίτες με τα διάφορα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, μπορούν οι πολίτες ε, να μαθαίνουν ποιες είναι αυτές οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται και προσπαθούμε να τα παρουσιάζουμε με τρόπο εύληπτο για αυτούς. Ε, όχι σε άμεση συνεργασία με τους πολίτες, αλλά ε, παρέχουμε προσανατολισμό, διότι δεν είμαστε εμείς ε, οργανισμός που απευθύνεται απευθεία στους πολίτες. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση και τις δημογραφικές αλλαγές, αυτό τέθηκε από πολλούς ομιλητές. Είναι προτεραιότητα για μας, αλλά οι επιπτώσεις δεν είναι πάντα σαφείς, διότι η δημογραφική αλλαγή ακόμη και σε ε, τομείς εργασίας που συρρυκνώνονται μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη δυναμικού. Γι' αυτό ε, εξετάζουμε διάφορα σενάρια. Εξετάζουμε, για παράδειγμα, αν η αυτοματοποίηση ε, έχει άμεσο αντίκτυπο στο σύνολο της δουλειάς ε, ή αν έχει επιπτώσεις εντός του χώρου αυτού, δηλαδή εάν μέρη της δουλειάς θα αυτοματοποιηθούν. Όσον αφορά τις χαμηλές δεξιότητες και τη δημογραφική αλλαγή, νομίζω ότι ήδη απάντησα στη... Ε, στην δημογραφική αλλαγή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, Υγείας Ε, δεν ε, ξέρω αν γνωρίζει τις εργασίες που κάνουμε εμείς. Και στον κύριο Άντζελ Αγχέλ, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς να προφέρω το όνομά σας, ε, ε, ε, επανακαθορισμός της κατανομής εργασίας. Καλό και τους άλλους αδερφικούς μας οργανισμούς να απαντήσουν στο θέμα αυτό. Δεν θα πρέπει να απαντάει μόνο ένας αδερφός. Νομίζω πάντως ότι υπάρχει διαφορετική εμπειρογνωσία εντός των οργανισμών μας, αλλά συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Κάποια παραδείγματα ήδη αναφέρθηκαν Έχουμε την κλασική συνεργασία ETF και SENDEFOP και να απαντήσω και εν μέρη και στο ερώτημα του κυρίου Βίλες. Ε, μπορεί να επικεντρωνόμαστε περισσότερο στις έρευνες ενώ ETF ε, είναι οργανισμός ε, εφαρμογής προγραμμάτων. Δοκιμάζουν λοιπόν τις διάφορες θεωρίες και μας αναφέρουν τα αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ε, ότι έχουμε σωστή ε, δομή. Ε, φυσικά μπορεί να υπάρξει επανακαθορισμός. Κάποια από τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε είναι κοινά και όλοι συμμετέχουμε στο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ναι πράγματι είναι πολύ σφιχτός και Ε, τέθηκε και άλλη ερώτηση. Πράγματι έχουμε αύξηση του φόρτου εργασίας. ο δικός μου οργανισμός τα τελευταία χρόνια ε, πρέπει να ε, καλύπτουμε περισσότερα θέματα, αλλά έχουμε ε, μειώσει κατά 10% το ε, αρχικό μας πρόγραμμα, τις αρχικές μας εργασίες, αλλά έχουμε και το, τη νέα αρμοδιότητα, το Central Market Intelligence. Από την άλλη δεν είστε εδώ για να γκρινιάξω ότι δεν έχω αρκετά χρήματα. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ε, βλέπουμε κάθε χρόνο πώς μπορούμε να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά και πώς μπορούμε να ε, κάνουμε καλύτερες έρευνες ε, χρησιμοποιώντας ε, το διαδίκτυο. Μπορούμε έτσι να εξοικονομήσουμε σημαντικά ποσά με τον τρόπο που διενεργούμε τις έρευνές μας. Ε, αλλά ναι, είναι σφιχτός ο προϋπολογισμός ε, και αν δούμε την νέα γενιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αν εξετάσετε τα έγγραφα αυτά, όλα έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες. Εμείς όμως ως ε, ΣΕΝΤΕΦΟΠ ε, είμαστε οργανισμός που τρέχει με μια σταθερή ταχύτητα. Αναμένεται λοιπόν ε, να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας με τον προϋπολογισμό που έχει προβλεφθεί για μας. Θα είναι δύσκολο αλλά θα το προσπαθήσουμε. Όσον αφορά τους τις εξωτερικές αναθέσεις. Νομίζω ότι το ποσοστό το δικό μας είναι κάπως λιγότερο από 30% γενικά θεωρώ προβληματικό το να έχουμε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ε, δύο κοινωνικές τάξεις, να το θέσω έτσι, αλλά δεν μπορώ εγώ να το λύσω. Όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση, νομίζω ότι ιδιαίτερα όσον αφορά τις έρευνες ε, είναι απαραίτητο να ε, κάνει κανείς εξωτερική ανάθεση, διότι αλλιώς ε, εμείς απλά θα ήμασταν κλεισμένοι στον, ε, στον όμορφο μας πύργο στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να βλέπουμε τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται εξωτερική ανάθεση κάποιων ερευνών. Κύριε Μίλλερ, όσον αφορά τις δεξιότητες, τις αλλαγές και πώς βρισκόμαστε σε επαφή με την αγορά εργασίας. Νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας, όπως εξήγησα και κατά τη διάρκεια της παρουσίασής μου. Βλέπουμε και πώς αλλάζουν οι δεξιότητες, πιστοποίηση ε, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την οικονομία των πλατφορμών που βλέπουμε. Ε, επίσης ε, οργανώνουμε φόρουμ ε, πολιτικής όπου καλούμε τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να δουν πώς άλλοι αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις. Υπάρχουν κενά, βρισκόμαστε κοντά στα όσα συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Όχι απολύτες, αλλά δεν είναι και αυτό το καθήκον μας. Είμαστε ευρωπαϊκός οργανισμός και σε πολλά κράτη-μέλη Υπάρχουν τοπικοί αδερφικοί οργανισμοί που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση στις διάφορες χώρες. Ε, από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να επιταχύνω. Ε, ε σας είπα πως ε, μοιραζόμαστε τα καθήκοντα με τη, τον ΣΕΝΤΕΦΟΜ και ETF. Κύριε Μπέκερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που έχετε αγκαλιά στον οργανισμό μας και για την υποστήριξη που μας υποσχεθήκατε. Με βρίσκεται απόλυτο σύμφωνο και να συνοψίσω τις ερωτήσεις που θέσατε, πώς ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη. Μαζί με το ETF συμμετέχουμε στη διαδικασία παρακολούθησης της ΡΙΓΑ και ε, όσον αφορά την κινητοποίηση εξετάζουμε και τα οικονομικά και μη οικονομικά κίνητρα ε, παρέχοντας προγράμματα άσκησης. Επίσης όσον αφορά το, το ΒΕΤ, την επαγγελματική κατάρτιση. Ε, επαναλαμβάνω την έκκλησή μας, ε, αν έχετε παιδιά, ε, σκεφτείτε να τα στείλετε να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση ως πρώτη επιλογή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να εστιάσω σε δύο. Η ψυχική υγεία και φίλο. Και μετά μπορώ να απαντήσω και κάποια πιο γενικόλογα. Πιο γενικά μάλλον ερωτήματα που αφορούσαν όλους τους οργανισμούς ε, για το φύλλο. Έκανε κάποιες ερωτήσεις και η κυρία Ρέγκνερ. Στο τομέα του φύλλου έχουμε κάνει πολλή δουλειά και θα έχουμε και τη στρατηγική για το φύλλο με ειδικά μέτρα για τη διαφάνεια στους μισθούς. Προσπάθησαμε να υπολογίσουμε το κόστος, για παράδειγμα, του μισθολογικού χάσματος, οι χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών, πάνω από το 2% σε σχέση, ε, μάλλον ποσοστό του ΑΕΠ. Βέβαια, με την αύξηση της απασχόλησης έχει αυξηθεί κάπως η απασχόληση των γυναικών, έχει, ε, και έχει μαθεί και το ποσοστό αυτό. Η Eurostat δημοσιοποιεί στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα. Εμείς προσπαθούμε να τηρήσουμε τις συστάσεις της Κομισιόν και βλέπουμε πώς εφαρμόζονται τα σχετικά σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των μισθών. Τι παίρνουν οι γυναίκες, τι παίρνουν οι άντρες. Και σε διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρεια. Οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν τις έχουν τηρήσει όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να λάβει υπόψη στις μελλοντικές σας συζητήσεις και τα αντισταθμίσματα. όταν έχουμε πιο μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας, η έκθεση ήταν ε, για κάστοτε πιο χρήσιμη. Αλλά δεν υπήρχε εξίσου μεγάλη συμμόρφωση γιατί ήταν δύσκολο. Άλλες χώρες ακολουθούν μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή γενικό λόγη. Προσέγγιση μεγαλύτερη συμμόρφωση, αλλά όχι τόσο μεγάλες λεπτομέρειες που μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρόσφατα έχουμε υπολογίσει το διοικητικό όκθος για τις επιχειρήσεις. Μας το ζήτησε DG, η ΓΔ Just. Και περιμένουμε σύντομα μια άλλη έκθεση, αυτή η κατέτοιμα της Κομισιόν. Συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φίλων, το ΕΙΓΕ, και δίνουμε στοιχεία για τον ε, ανάλογο ε, δίκτυ της ισότητας των φύλων. Εσωτερική διαχείριση στο Eurofound έχει τους στόχους της. Ε, μια άλλη συνάδελφο ε, που έκανε στα ισπανικά τι ερωτήσει, τη, θα μπορούσα λοιπόν να τι απαντήσω εγώ στα ισπανικά. Βάλτε λοιπόν παρακαλώ τα ακουστικά σα. Ναι, πράγματι, συμμερίζομαι την ανησυχία σας για την ψυχική υγεία και την ε, ψυχική υγεία και ευεξία των εργαζομένων. Εμείς ε, ασχολούμαστε πολύ και έχουμε και πέντε ένα δείκτη πέντε στοιχείων από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Προσπαθούμε να συσχετίσουμε τα στοιχεία για να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες εργασίες που φέρνουν καλύτερη ψυχική υγεία και ευεξία. Φέτος έχουμε την επιτόπου εργασία για τη νέα έρευνα για την απασχόληση. Πάνω από 42.000 εργαζόμενους στα ε, έχουμε ρωτήσει με συνεντεύξει όπως είπα και είμαστε σε επαφή επίσης ε, με την Όσα και τον αδελφό φορέα γιατί πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία της έρευνας για να βάλουμε σε ένα πλαίσιο και να ερμηνεύσουμε αυτά τα στοιχεία. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, καταλαβαίνετε, γι' αυτό συνεργαζόμαστε με τους οργανισμούς. Επίσης, ε, βλέπουμε η ψηφιοποίηση τι αντίκτυπο μπορεί να έχει σε ό,τι αφορά τα περισσότερα βάρη το, εργα... το, το άχθος. Επίσης το δικαίωμα στην αποσύνδεση, ρύθμιση και κοινωνικές συμφωνίες. Είναι κάτι που επίσης μας ενδιαφέρει, το έχουμε ήδη κάνει και θα έχουμε τη σχετική έκδοση τον Απρίλιο. Και να ξαναμιλήσω αγγλικά για κάποιες γενικές καταληπτικές παρατηρήσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη Βερόνικα Λόπεθ Φαντανιέ Muchas gracias. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πολύ μιλήσατε για τον προπολογισμό. Να ευχαριστήσω τον Αλεχάνδρο Θέρκας. Gracias. Έχουμε υψηλές προσδοκίες και υψηλές απαιτήσεις από το ΔΣ και τους άλλους ε, πρώτης αρχής γενομένης από την Κομισιόν αλλά και όλων των άλλων εμπλεκομένων. Αν δείτε τις εκτιμήσεις ε, για την επταετία του ΠΔΠ, εμείς θέλουμε να προωθήσουμε τις έρευνες για να δούμε αν είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Πρέπει να διατηρηθούν. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Το συζητούμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές όταν ε, θέτω αυτά τα στήματα μου λένε «Α, θα υπάρξουν ε, <clears throat> κάποιες ανάγκες ε, προσαρμογής και θα τα καταφέρετε». Ήδη έχουμε μειώσει 10% το προσωπικό, έχουμε μειώσει τον προπολογισμό σε πραγματικούς όρους. Λαμβάνουμε υπόψη το βετικό επίπεδο στην Ιρλανδία και τους μισθούς. Άρα όλο και μειώνονται τα ποσά. Και γι' αυτό, όπω είπατε και εσεί κύριε εμεί θέλουμε να εξερμίσουμε όλε τι δυνατέ επιλογέ για συνέργειε. Το θέμα είναι βέβαια να αποφασιστεί όχι από εμά, γιατί δεν είναι δική μα αρμοδιότητα, πόσοι οργανισμοί πρέπει να έχουν για ποιο θέμα και όταν αυτό έχει καθοριστεί πλέον θα δούμε τι θα κάνουμε, θα υπάρξει συνεργασία. Πρέπει χάρη όπω έχουμε ε, στο front office, αν θέλετε, με τι επιχειρήσει ή back office ε, με σε άλλους τομείς. Έχουμε το δίκτυο ευρωπαϊκών ε, γασμών και άλλα. Αλλά επειδή είμαστε ξεχωριστές νομικές οντότητες, ε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο καλά ε, αυτή η συνέργεια. Αν υπάρχει μια δομική νομική βάση, μπορούμε να το κάνουμε. Για κοινέ υπηρεσίε, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κοινέ υπηρεσίε. Όλοι όμω προ εκεί προσδοκούμε να πάμε και έχουμε το μνημόνιο συνεννόησης. Τα προγράμματα εργασία μα είναι γνωστά σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψει και αντίθετα να εντοπίζονται και δυνατότητε συνέργεια σε πολύ ε, πρόωρο στάδιο, ακόμα και πριν δημοσιοποιηθεί το πρόγραμμα εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, κυρία Σέντλατσοκ, γιατί αποδεικνύουν ότι ενδιαφέρεστε για το θέμα. Και το ενδιαφέρον σας είναι κίνητρο για μένα και για τους συνεργάτες μας. Μιλήσατε για επικίνδυνες ουσίες και τα καρκινογόνα. Ναι, όντως είναι προτεραιότητά μας. Διαπνέει τις δραστηριότητές μας, τα προγράμματά μας. Οπότε αυτό πρέπει να τονίσετε. Πρόκειται για το ανθρώπινο δικαίωμα στην ασφάλεια για να δούμε όμως ποιο είναι το κόστος αυτών των ε, ασθενειών που έχουν πήγει τον εργασιακό χώρο. Πόσα δις ευρώ δαπανώνται από τις ε, εταιρείε και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στην εργασία. για να δούμε επομένω, τι σημαίνει να μην λαμβάνονται τα μέτρα κατά των ε, καρκινογόνων και επικινδύνων ουσιών. Βεβαίω και θα συνεχίσουμε την καμπάνια μας για υγεία στον χώρο της εργασίας. Βεβαίω και θα παρουσιάσουμε την επιστημονική τεκμηρίωση που υπάρχει και σε πολλά επίπεδα αυτό πρώτα-πρώτα πρακτικές, ε, πρακτικά παραδείγματα από εταιρείε. Ακόμα και σε μικροεταιρείες, μικροεπιχειρήσεις είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα. Μέτρα τα οποία να μην κοστίζουν και τόσο πολύ. Γιατί με τις εταιρείες που συμμετέχουν στην προστασία μας θα αναδείξουμε το τι ισχύει με μειοσκελετικές ασθένειες κλπ. Και με προβολή των καλών πρακτικών να καταδείξουμε ότι είναι δυνατή μία αντιμετώπιση. Σε πολλά μετωπιμένες είδαμε ότι η κινητοποίηση και τα κίνητρα τα καλύτερα προέρχονται από άρτια νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι το μέσο για να αναβαθμιστεί η ασφάλεια του χωροεργασία. εργασίας. Στην προηγούμενη θητεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσπαθήσει για αυτές τις ουσίες να τροποποιήσει την νομοθεσία και ο Επίτροπος Σμιτ πρόκειται να συνεχίσει αυτό το έργο. Τα γενετικά τροποποιημένα, τα καρκινογόνα κλπ. Τώρα, σε σχέση με κάτι άλλο. Έχουμε διάφορους ε, παράγοντες σε σχέση με τις επικοινωνικές ουσίες, ε, όπως σας πούμε αναφερθήκε η νυχτερινή βάρια, η νυχτερινή εργασία, βεβαίως και έχουμε έρευνες που κατατείνουν στο ότι υπάρχουν επιπτώσεις, ότι επηρεάζει το ένα το άλλο. Οπότε και φέτος αρχίσαμε να εξετάζουμε τι γίνεται με την έκθεση του εργαζομένου σε καρκινογόνα. Νέα μεθοδολογία. Έτσι θα διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες στο χώρο εργασία, σε συγκεκριμένους τομείς που επηρεάζουν. Και θα καλύψουμε και την εργασία τη νύχτα. Άρα να δούμε πώς συνδυάζονται διάφοροι παράγοντες που όλοι μαζί σχετίζονται με τον καρκίνο τώρα ψυχοκοινωνικός κίνδυνος. Και αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα γιατί είδαμε αύξηση εργασιακών ασθενειών σε σχέση με ψυχοκοινωνικές ε, παθήσεις. Και βέβαια και η διανοητική ψυχική υγεία έχει σχέση και με τις νέες δραστηριότητες όπως τα ψηφιακά. Να καταλάβουμε τι σημαίνει κανείς να δουλεύει σε μια πλατφόρμα ή να δουλεύει με ρομπότ. Ακόμα είναι μικρή η εμπειρία μας. Όμως, αυτό θα είναι κομμάτι της προσπαθειάς μας. Κάπου να καταλήξουμε και να διατυπώσουμε και κάποιες ε, συστάσεις. Γιατί υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες μεγάλες εταιρείες που έχουν καλές πρακτικές. Για την ψηφιοποίηση βέβαια. Θα συνεργαστούμε με τις άλλες υπηρεσίες για να δούμε πώς επηρεάζουν. Επίσης, η ψηφιοποίηση έχει σχέση, είπαμε, ε, με τις μυοσκελτικές ασθένειες και αυτό θα είναι το αντικείμενο της νέας καμπάνιας. Επανέρχομαι τώρα. Α, για δούμε πρώτα στα θέματα ισότητας των φύλων. Είναι οριζόντιο το ζήτημα. Προσπαθούμε εμείς να το εντάξουμε σε όλε τι δραστηριότητε μας. Και τις επικοινωνίες ουσίες επίσης. Υπάρχουν ε, σαφή ευρήματα ότι σε κάθε φύλλον διαφορετική επίδραση των επικίνδυνων ουσιών. Οπότε χρειάζονται και διαφορετικά μέτρα. Και τα μειοσκελετικά είπαμε. Υπάρχει θέμα στον ε, κλάδο υπάρχει υπηρεσιών. Αυτές οι ασθένειες είναι κάτι ε, το οποίο είναι αποτέλεσμα του ρίσκου του κινδύνου αυτού του κλάδου. Οι προηγούμενοι συνάδελφοι είπαν ότι ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί περικοπές για την επόμενη περίοδο, για την επόμενη χρονιά. Εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε τη δραστηριότητά μας, τη των άλλων υπηρεσιών και έτσι να οργανωθούμε. Άρα αυτό είναι μόνιμη μέρη μας μας αποσχολεί όλους και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε μέσα στην εντολή μας κάτι να κάνουμε. Καλά, πέστε μου αν ε, κάτι ξέχασα. Η πρόεδρος. Κοιτώ δεξιά-αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τι ερωτήσει σας ε, προς το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματική εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω από το φόρτο εργασίας και τον προϋπολογισμό. Έτσι ξεκίνησε η νέα στρατηγική. Έπρεπε να εργαστούμε με βάση τις προτάσεις που ήδη υπήρχαν. Προϋπόθεση ήταν λοιπόν να παραμείνει ο προϋπολογισμός σταθερός, ε, μη λαμβάνοντας υπόψη τον, τον ε, πληθωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει επηρεάσει την ε, διαφοροποίηση και τη στόχευση στις εργασίες μας. Και καθώς και την εξέβρεση συνεργειών με δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως γενικά ε, στις ε, ε, εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξωτερική δράση όσον αφορά τις δεξιότητες κτλ. Δεν υπάρχει έλλειψη πόρων. Αυξάνεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητε και τις, τις δεξιότητες και την επαγγελματική κατάρτιση. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε ακριβώς στις εργασίες αυτές, ε, πετυχαίνοντα έτσι, την καλύτερη δυνατή συνέργεια. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε με διάφορους εταίρους ε, και συνομιλητές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Γενικές Διευθύνσεις, ΔΕΦΚΟ, ΝΙΕΡ κλπ. Ακούσατε διάφορες απόψεις. Εμείς εργαζόμαστε εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, ωφελούμαστε από την ανταλλαγή απόψεων και εμπειρογνωσία με τους άλλους συναδέλφους μας, ιδιαίτερα την Eurofound καθώς ε, και τον ΣΕΝΤΕΦΟΠ σε διάφορους τομείς. Ε, δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη ανέφερε ο Γιούργεν. Όσον αφορά τις, τις δεξιότητες στο μέλλον στις μεσογειακές χώρες. Ε, έχουμε τη διαδικασία του Τωρίνο. Θα πάμε λοιπόν φέτος στις ε, χώρες ε, της Μεσογείου. Είχαμε μεγάλη διεθνή διάσκεψη πριν δύο χρόνια που εξετάσαμε ιδιαίτερα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στις χώρες εταίρους μας. Και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διαφορά, υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που έχουν γίνει γνωστά για τη ρομποτοποίηση, την ε, ε, βιομηχανία 2.0, ε, την ε, διάγνωση του Νταβός και την πραγματικότητα σε πολλές από τις χώρες εταίρους μας, όπου αυτά ισχύουν για πολύ μικρό μέρος της οικονομίας. Ενώ γίνεται λιγότερη δουλειά πάνω στις παραδοσιακούς τομείς που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά, πώς ε, μπορούμε να δούμε πού υπάρχουν αναντιστοιχίες ε, στις ε, θέσεις εργασίας και να εξετάσουμε τους διάφορους τομείς. Την πρώτη τομεακή μελέτη θα την έχουμε μέσα του 2020 και με αυτήν ως βάση θα αναπτύξουμε συστάσεις και θα μοιραστούμε τις ιδέες μας με τις γειτονικές μας χώρες. Αυτός λοιπόν είναι σημαντικός ε, τομέα δουλειά, Σας ευχαριστώ πολύ που το αναφέρατε όσον αφορά τις δεξιότητες, τη θεωρία και την πράξη. Εμείς εργαζόμαστε σε πρακτικό επίπεδο. Μάλιστα, αποφελούμαστε από πολλές από τις έρευνες που γίνονται από τον ΣΕΝΤΕΦΟΠ και άλλους φορείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οποίους ε, στηρίζουμε τη σειρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Είναι πολύτιμη η εμπειρογνωσία στα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά στις ε, χώρες εταίρους μας. ενδιαφέρον παράγοντας όσον αφορά τον τρόπο εργασίας μας είναι ότι είναι πολύ πρόθυμοι οι ε, εταίροι μας. Ενώ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι εθνικές αρμοδιότητες. Ενώ στα, στο πλαίσιο συνεργασίας με τρίτους ε, μπορούμε να συνεργαστούμε με εταίρους που επωφελούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα ε, των δεξιοτήτων και των ωφελών. Ε, έχουμε μια διάσκεψη τον έμβριο για τις δεξιότητες και εξετάζουμε το όφελος ε, για τους ανθρώπους, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά παραδειγμάτων καλών πρακτικών σε διάφορες περιοχές, μεταξύ άλλων τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συλλέξει εκατοντάδες παραδείγματα και έχουμε εκπονήσει εγχειρίδιο σχετικά με το πόσο μπορούμε να ε, ε, ενσωματώσουμε την πτυχή αυτή, ε, να εξετάσουμε και τις νέες μορφές οικονομίας, την οικονομία της πλατφόρμας και άλλα. Όσον αφορά τα οριζόντια θέματα που μας ρωτήσατε σχετικά με, τα, με την ισότητα των δύο φύλων και τη δημογραφία, δεν θα προσθέσω πολλά σε τα όσα υπόθηκαν. Είναι σημαντική πτυχή όταν συζητάμε την αλλαγή των συστημάτων ε, στα κρατημέλη. Αυτοί είναι σημαντικοί πυλώνες ε, κατά την ανάλυση και την εκπόνηση προτάσεων ε, προς τις χώρες αυτές. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους διάφορους τομείς. Κάποιες από τις χώρες μας έχουν ε, δημογραφικές εξελίξεις και ισότητα που να αντικατοπτρίζουν λίγο πολύ την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν σημαντικές αλλαγές. Όσον αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είναι χαρά μου να σας ε, ανακοινώσω ότι έχουμε περισσότερες γυναίκες. Έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον εργασίας που το αντικατοπτρίζει αυτό και το Διευθυντικό Συμβούλιο είναι ισορροπημένο όσον αφορά τα δύο φύλλα. όσον αφορά τα θέματα που έδειξαν οι παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τους ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις τους και ε, την ενθάρρυνσή τους. Ε, σας ευχαριστούμε για την υψηλή ποιότητα των ε, συνεισφορών σας, διότι αυτό είναι που καθορίζει και την εμπειρογνωσία μας πολύ σωστά. Τονίσατε το θέμα της φιλοδοξίας, την τους στόχους μας σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συνεχώς. Και έχουμε δημιουργήσει μια προσέγγιση με τη νέα στρατηγική, η οποία να μην εμποδίζει την ε, συνέχιση της διεξαγωγής αυτής της συζήτησης. Έχουμε 19 χώρες εταίρους, ε, τις χώρες ε, γειτονίας. Έχουμε περιορισμένους πόρους, είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε περαιτέρω στις εργασίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έξω από τις χώρες εταίρους αυτές, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει με τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, μπορούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα με τους πόρους που έχουμε εντός της εντολής που έχουμε. Αν όμως ε, θέλουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, θα πρέπει να θέσουμε το θέμα των ε, διαθέσιμων πόρων. Ε, λαμβάνω γνώση των ε, παρατηρήσεων του κυρίου Σέρκας αλλά και του κυρίου Μπάουερ σχετικά με το αν θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ε, σχέσεις με την Επιτροπή ΔΕΒΕ ή και με άλλους. Η δομή του οργανισμού μας αντικατοπτρίζει τον τρόπο διαχείρισης από πλευράς της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργαζόμαστε και με τους άλλους παρόντες οργανισμούς αλλά ασχολούμαστε και με την διάσταση των εξωτερικών σχέσεων. Ίσως ε, θα έπρεπε να ε, υιοθετήσουμε την πρότασή σας και να επικεντρωθούμε περισσότερο στις ε, προτάσεις συνδυασμού της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης. στις δικές μας σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, η Γενική Διεύθυνση ΝΙΕΡ και η ΕΙΕΔ είναι οι συνομιλητές μας για πολλά από τα θέματα που έχουμε μπροστά μας. Αναφερθήκατε και στην Αφρικανική Ένωση και εδώ μπορεί να υπάρξουν δυνατότητες ανάπτυξης. Συνεργαζόμαστε όσον αφορά ε, το ε, ε, πλαίσιο δεξιοτήτων του συνόλου της Αφρικής. Ε, το ETF, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ε, συμβάλλει με την εμπειρογνωσία του. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Έλα για τις τελευταίες παρατηρήσεις. Εγώ θα πάρα πολύ σύντομο γιατί δύο ερωτήματα αφορούσαν τη δική μας υπηρεσία. Το ένα ερώτημα ήταν το των επιθεωρήσεων. Όπως είπα, θα είναι πάνω από μία όπως ζητήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό θα πράξουμε και να πω και αυτές εξ ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχουν πολλές διμερεί συμφωνίε. μεταξύ εθνικών επιθεωρήσεων εργασία στην Ευρώπη. Θα επιβλέπουν αυτές τις τονισμένες δράσεις. Εμείς, ε, επομένως, ε, αυτό που θα κάνουμε είναι να δώσουμε μορφότυπα και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν αυτοί που θα αναλάβουν αυτές τις επιθεωρήσεις ως επιπρόσθετη συνδρομή, όχι αντικαθιστώντας κάτι που ήδη υπάρχει. Και το δεύτερο ερώτημα, το κατά πόσον έχουμε ήδη επιληφθεί θεμάτων, ε, κοινωνικούς εταίρους κτλ. Από την ΕΤΟΚ έχουμε ενημερωθεί με επιστολές για διάφορες ε, υποθέσεις που αφορούν δύο περισσότερα κρατημέλη, για την απόσπαση των εργαζομένων πράγματι, ήταν πολλά από αυτά τα θέματα, κακές συνθήκες εργασίας από τον απόσπασμένο εργαζόμενο κτλ. Και έχουμε και την εφαρμογή του άρθρου 8. Δηλαδή, στέλνουν αυτές τις επιστολές στα μέλη του ΔΣ που εκπροσωπεί το κάθε κράτος. Εγώ τώρα συλλέγω τις απαντήσεις τους για να ενημερώσω τους κοινωνικούς εταίρους. Στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε όλα τα άρθρα του κανονισμού και το 8 επομένως, εξού και θα προβλεφθεί ειδική διαδικασία είναι ένα θέμα σημαντικό. Απ' την άλλη, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στις επιθεωρήσεις διαφέρει από κράτος μέλος σε, κάτω, σε κράτος μέλος. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος ρόλος, σε άλλες κράτη όχι. Αυτό το γνωρίζουμε. Το ξέρουν και τα μέλη του ΔΣ. Θα βρούμε λοιπόν το πιο ενδεδειγμένο σενάριο για την κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και μας παρουσιάσατε το πρόγραμμα εργασία και το έργο που έχετε επιτελέσει και θα επιτελέσετε. Ευχαριστώ και τους ε, εισηγητέ που ήρθατε στην Επιτροπή. Νομίζω ότι έχουμε ε, αποκομίσει μια πολύ πληρικό. Να συνεχίσετε την καλή δουλειά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα ήθελα τώρα να αφήσω την θέση της Προέδρου σε ένα μέλος του Προεδρείου. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Bom dia a todos. Vamos continuar os trabalhos desta sessão da manhã. Καλημέρα και από πλευρά μου, λέει η πρόεδρο. Ε, συνεχίζουμε την ε, ημερήσια διάταξη με το επόμενο σημείο που είναι η παρουσίαση τη έκταση του Eurofund με θέμα τη σύνθεση και την ευημερία των οικοκυριών. Έστερ Σάντορ είναι η προσκεκλημένη μα. Ε, θα μα παρουσιάσει την έκταση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τότε. Σα παρουσιάσω αυτό το πόνημα το είπε και ο Χουάν ότι έγινε αυτή η έρευνα και την Ελεονόρα που θέλω να την ευχαριστήσω που συνεργαστήκαμε για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Είναι μια έκθεση η οποία θέλει να παράσχει μια εικόνα για τη σύνθεση των οικοκυρών στην Ευρώπη και να παρουσιάσει τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία Θέλαμε να ελέγξουμε μήπως υπάρχουν κάποια νοικοκυριά τα οποία είναι παραμελημένα λόγω των πολιτικών κρατών μελών ή κάποια μέλη των νοικοκυριών, μήπως αφήνονται εκτός. Δεν ασχολούνται τα κράτη-μέλη με τις πολιτικές τους. Χρησιμοποίησαμε τα διατομεακά στοιχεία και στη, στηριχτήκαμε στη δεκαετία 2017 και για την ευημερία συγκρίναμε τις χρονιές 2007 και 2016 ε, την Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής. Είδαμε ανάδειξη οικογένειες ε, και μελετήσαμε και την ε, των παιδιών. Ποια είναι τα βασικά είδη νοικοκυριών. Μόνο πρόσωπα νοικοκυριά, ζευγάρια, κυρίως τη συμβίωση, συγκατοίκηση και όχι τα έγγαμα ζευγάρια, ζεύγη με παιδιά, ομοφυλόφιλα ζευγάρια και συνταξιούχους. Είδαμε το τρίτο ε, νοικοκυριά με παιδιά, μονογονικές οικογένειες, ε, ανάδοχες ε, και βασικές οικογένειες και τέταρτον είδαμε πολυγενειακά νοικοκυριά, νέους που ζουν τους γονείς τους, ε, μεγάλα και πολύπλοκα δηλαδή νοικοκυριά για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Ένα τρίτο των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μονοπρόσωπα. Και πρέπει να τους δοθεί προσοχή γιατί υπάρχει αύξηση αυτό του ποσοστού σε όλες τις χώρες σχεδόν στην Ευρώπη. Υπάρχει μόνο μια πηγή εισοδήματο, ε, γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχεια για αυτά τα νοικοκυριά. Σε κάποιες χώρες η αναλογία αυτή είναι μεγαλύτερη στην Ανατολική Ευρώπη, Βουλγαρία, Μαγκαρία Υπήρχαν χώρες που είχαν τα υψηλότερα ποσοστά, Δανία, Βέλγιο, Φιλανδία, Σουηδία μεταξύ άλλων, που υπάρχει πλέον μείωση σιγά σιγά. Ηλικίες επίσης. Στην Ανατολική Ευρώπη οι νέοι είναι πιο ηλικιωμένοι και όχι νέοι. Έχουν χάσει τον σύντροφό τους έχει αυξηθεί και το προσδόκιμο επιβίωσης. Άρα οι γυναίκες πιο πολύ ζουν μόνες τους. Οι νέοι επίσης ε, όλο και περισσότερο, οι άντρες οι γυναίκες μένουν μόνοι τους γιατί δεν μπορούν να ζήσουν πλέον στο, στην οικογένειά τους. Στις βαλτικές χώρες έχουμε το μεγαλύτερο ε, κίνδυνο φτώχειας και ο μικρότερος είναι η Ισπανία, Ουγγαρία, Ελλάδα. Έχω και κάποια για την υγεία στην έκθεση για όλε τι ηλικίε ομάδε. Η υγεία, όπω την αναφέρουν οι ίδιοι, είναι χειρότερη για αυτούς που ζουν μόνοι του. Όχι μόνο για του πιο ηλικιωμένου. Όλοι το λένε αυτό. Οι μεγάλοι όλο και περισσότερο βέβαια. Στην Κροατία είχαμε τη μεγαλύτερη αναλογία ηλικιωμένων στη μελέτη ε, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά με κακή υγεία. Ιρλανδία 8% μόνο α, για τι ηλικίε άνω των 65, που έλεγαν ότι δεν έχουν καλή υγεία. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτοί που ζουν μόνοι του χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο και τι υπηρεσίε υγεία. Προσπαθώ να τα πω πάρα πολύ γρήγορα για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Ευτυχία. Από ένα στα δέκα όσοι μένουν μόνοι τους είναι λιγότερο ευτυχείς από αυτούς που ζουν με άλλους. Στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ μεγάλο το χάσμα και σε κάποιες ε, χώρες της Ευρώπης όπως την Πορτογαλία. Που μπορεί όμως βέβαια να οφείλεται και στο ότι δεν είναι επιλογή αλλά αποτέλεσμα το τέχασμα των συντροφών του το να μένουν μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι. Για τις μεσαίε ηλικίε ομάδε, τα 65 και 60 εκεί βλέπουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά. Ίσως γιατί είναι και πιο ασυνήθιση ηλικία για να είναι κανείς μόνος του και να ζει μόνος του. Αν δεν υπάρχουν επαρκείς κοινωνικές επαφές, αυξάνεται η αίσθηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η αίσθηση της ε, δυστυχίας. Ε, Σημειώσαμε επίσης επίσης ότι υπάρχει παρόλα αυτά ε, μεγαλύτερη ευτυχία για όσους ζουν ε, ανεξάρτητοι από το να ζουν σε σχήματα ε, πολύπλοκα. και επίσης και η ψηφιακή συνοχή ως σημαντικό ζήτημα. Um, Για τα ζευγάρια τώρα το 1 τέταρτο των οικοκυριών. Δύο άτομα δηλαδή σε σχέση. Είδαμε τις κατοικίες καταρχάς έναντι των έγγαμων ζευγαριών. Γιατί είδαμε τις κατοικήσεις, γιατί αυξάνουν τα ποσοστά σε όλες σχεδόν τις χώρες αυτή τη δεκαετία που μελετήσαμε. Και δυστυχώ όσοι συμβούν δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με του έγγαμου σε περιπτώσει. Στη Γαλλία και στι βόρειε χώρε. Πολλά ζευγάρια μένουν πολλά χρόνια μαζί πριν παντρευτούν και παντρεύονται πολλές φορές μετά το πρώτο παιδί. Αλλά αυξάνεται και στις άλλες χώρες. Στη Βουλγαρία μετά το 7 και στην Εστονία είδαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Σε ό,τι αφορά την ευεξία και την καλή κατάσταση. Υπάρχουν δικαιώματα πλέον ε, χαμηλότερες, ε, χαμηλότερα φόρο, φοροϊκά κίνητρα, χαμηλότερη φορολογία, κάποια δικαιώματα και επιδόματα που παίρνουν και έτσι αυτό βελτιώνει κάπως την κατάσταση παρά το γεγονός ότι αυτά τα ζευγάρια μπορούν να μπαντρεύονται αμέσως ομοφυλόφιλα ζευγάρια να πω, και ομόφυλα ζευγάρια να πω κάποια πράγματα. Δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Θέλαμε να δούμε κατά πόσο εκπροσωπούνται σε επίσημε στατικέ και έρευνε και καταλήγουμε στο εξή συμπέρασμα. Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα στην, ε, σε σχέση σχέσεις ή που εκπροσωπούνται αυτά τα ζευγάρια. Έχουμε μικρό δείγμα λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το εισόδημα, τη στέγαση, τα πράγματα είναι παρόμοια. Αλλά κυρίως στον κοινωνικό αποκλεισμό και την χαμηλότερη στήριξη από την οικογένεια, εκεί βλέπουμε διαφορά στα ποσοστά. Άρα βοηθάει η κοινωνική υποστήριξη και μειώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Uh, Retired uh, συνταξιούχοι. Αυξάνεται λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής ιδίως για τους άνδρες. Και έτσι έχουν περισσότερα ε, νοικοκυριά που απαρτίζονται από δύο συνταξιούχους. Βλέπετε τα ποσοστά. Μετά την ηλικία των 65. Η ευεξία είναι πολύ μεγάλη αν κανείς ζει με το σύντροφο ή τη σύντροφό του. Αυτό επίσης δεν έχει οικονομικά ωφέλη. Υπάρχει έντονη πτυχή φίλου Οι γυναίκες είναι περισσότερο από τη φτώχεια. 37% λιγότερο παίρνουν ως σύνταξη γυναίκες. Οι γυναίκες που δεν παντρεύτηκαν ή που έχουν χωρίσει και αυτές που έχουν χειρέψει κινδυνεύουν περισσότερο να μην σε κάτω από το κατόφλι της στόχιας. Νοικοκυριά με παιδιά. Είδαμε καταρχάς τις οικογένειε χωρίς παιδιά. Γιατί αργούν να γεννήσουν οι γυναίκες πολλές φορές. Άρα θα αυξηθεί και αυτή η κατηγορία. Αλλά δεν είχαμε μεγάλη αύξηση σε άτεκνα ζευγάρια στην Ευρώπη. Στι Βαλτικέ είχαμε μια ελαφρά αύξηση αυτών των ζευγαριών. Τώρα σε αυτές ε, τις ε, οικογένειε ε, που είναι βασικέ, α πούμε, στοιχειώδη πυρήνα γονείς και παιδιά είναι 25%. Στην Κύπρο, στη Λιθουανία, στη Λετωνία, στη Μάλτα και στην Ουγγαρία μειώνουν τα ποσοστά. Λόγω το ότι αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και τα πιο ηλικιωμένα βαριά σε Ελλάδα και Ιρλανδία. Όμω είναι η βασική μορφή οικογένεια ακόμη, το βασικό νοικοκυριό. Αν συγκρίνουμε άτεκνα και μη ζευγάρια, ενώ μπορεί να υπάρχουν κάποια άλλου είδους ωφέλη για τα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά οικονομικού είδους κτλ. Η ευτυχία είναι μεγαλύτερη στα ζευγάρια που έχουν παιδιά. Και πολλές φορές υπάρχουν δύο εισοδήματα, γιατί είναι τα ζευγάρια νέα. Οι πατεράτες με παιδιά εργάζονται πιο πολύ από αυτούς που δεν έχουν. Και έχουν μεγαλύτερο στρες. ογκαρια Βέλγιο. Μεγαλύτερες διαφορές. Οι μητέρες τώρα μπορούν μάλλον κάνουν περισσότερη οικιακή εργασία, ακόμη και αν εργάζονται, πάνω από τις μισές. Έως 14 περισσότερες ώρες την ημέρα στο σπίτι, συν των άλλων υποχρεώσεών τους. Δηλαδή, αν δουλεύουν, έχουν και να φροντίσουν. όπως σας είχα πει και αλλού. Και αυτά βέβαια ε, συμβάλλουν στο να είναι χαμηλό το εισόδημα. Έχουν δείξει διάφορες έρευνες ότι η ε, επένδυση σε εκπαίδευση πολύ μικρών παιδιών ε, καθώς ε, και σε προγράμματα που βοηθούν τους άντρες και τις γυναίκες να μοιράζονται καλύτερα το φόρτο συμβάλλουν καλύτερα σε καλύτερη ισορροπία οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Εδώ έχουμε τα μονογονεϊκά νοικοκυριά. τα περισσότερα προγράμματα σκοπό έχουν να επαναφέρουν στην εργασία ε, τους ε, μόνους γονείς. Ε, είδαμε αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη, στα νοικοκυριά αυτά. Σε κάποιες χώρες είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση, ενώ σε άλλες όχι τόση. Η έκθεσή μας ε, δείχνει ότι μπορεί να ε, βελτιωθεί η κατάσταση για τα νοικοκυριά αυτά. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ε, ένα παράδειγμα όπου λαμβάνουν επιδότηση εισοδήματος και ενθαρρύνονται στην εξέβρεση εργασίας, αλλά αυτό αυξάνει την πίεση στους γονείς αυτούς πιο πιθανό να βελτιώσει την κατάσταση των οικοκυριών αυτών είναι η επένδυση σε δομές φροντίδας των παιδιών. Μικτές οικογένειες, ε, εδώ υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τους τύπους νοικοκυριών. Υπάρχουν στοιχεία ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός τους και έχουμε όλο και πιο πολύπλοκες δομές, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να τις καλύψουμε με επίσημες στατιστικές. Αλλά τα διαζύγια είναι πιο συνηθισμένα τώρα από ό,τι ήταν ε, παλιά και πολύ συχνά τα ε, παιδιά ε, μένουν ε, μια στον έναν γονέα, μια στον άλλον. δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, υπάρχουν όμως κάποια ε, δεδομένα και φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση στις χώρες όπου υπάρχουν στατιστικές, στην Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες. Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την ε, Ποιότητα Ζωής ε, δείχνει ότι γενικά βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση αυτές οι οικογένειες παρότι είναι και μεγαλύτερης ηλικίας από ότι οι μόνοι γονείς έχουν συζητηθεί οι διάφορες οικογενειακές ρυθμίσεις σε κάποιες χώρες. Οι έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η αναγνώριση ε, του καθεστώτος των ε, πατριών και μητριών ε, βελτιώνει και την ευημερία των παιδιών. Τέλος, έχουμε κάποια πιο μεγάλα και πιο πολύπλοκα νοικοκυριά, νοικοκυριά με περισσότερες γενιές. Ε, αυτό σημαίνει τρεις ε, γενιές τουλάχιστον, ε, δηλαδή παππούδες, γονείς και παιδιά. Οι γονείς και παππούδες που ζουν σε τέτοια νοικοκυριά βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από τις άλλες οικογένειες και φαίνεται ότι όταν τρεις γενιές ζουν μαζί αυτό η περισσότερο είναι ανάγκη ε, λόγω ανάγκης φροντίδας ή λόγω περιορισμένου εισοδήματος. οι γονεί ε, στα νοικοκυριά αυτά ε, συνήθως δεν χρειάζεται να φροντίσουν τόσο πολύ τα παιδιά διότι αυτό το, το φροντίζουν οι παππούδε. αλλά ε, απ' την άλλη πρέπει να φροντίσουν του παππούδε. και οι μεγαλύτερε διαφορές στην ευημερία ήταν σε αστικές περιοχές, στις υπαίθριες περιοχές δεν ήταν τόσο μεγάλε οι διαφορέ. Τα παιδιά πάντως δεν επηρεάζονται αρνητικά, αντιθέτως επωφελούνται από την παρουσία των παππούδων. Και το τελευταίο είδος νοικοκύριου που θα αναφέρω είναι οι νέοι ενήλικες που ζουν με τους γονείς τους, αυξάνεται το φαινόμενο αυτό. Ε, και αυτό δεν συμβαίνει απαραίτητα λόγω της κρίσης Η αύξηση ήταν κυρίως για τις νέες γυναίκες ε, μέχρι ηλικίας 24 ετών ε, που είναι πιο πιθανό να ε, σπουδάζουν αντί να παντρεύονται. Τα συμπεράσματα λοιπόν, η αναγνώριση των διαφόρων μορφών οικογενειών στην κοινωνική πολιτική μπορεί να βελτιώσει την ευημερία στα νοικοκυριά. η αναγνώριση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερα προβλήματα ε, ε, και διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα σε μεγαλύτερες ε, ηλικίε. Είναι σημαντικό να διευκολυνθούν οι, άδειες, οι γονικές άδειες των παιδιών και πρέπει να υπάρχει και κοινωνική υποστήριξη πέρα από, τα, από τις οικονομικές επιδοτήσεις για μονογενεϊκές οικογένειες. Αυτά είχα να πω. Ζητώ συγγνώμη ε, που τα είπα γρήγορα. Ελπίζω να μπορέσω να σας δείξω πόσο σημαντικές είναι αυτές οι έρευνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, ευρωβουλευτές. Μας είπατε αυτούς της ευπαθείς ευάλωτες ομάδες και τις σχετικές πολιτικές που πρέπει να δημορφωθούν Τώρα για πέστε μας με τα οικοκυριά που δεν εμπλέκουν οικογένεια. Τι γίνεται για τη στέγαση και τα πάνε εκεί ακριβένουν. Τι γίνεται, όλο ένα και περισσότεροι μένουν μαζί, μοιράζονται ένα διαμέρισμα. Εσείς θεωρείτε ότι θα υπάρξει αύξηση ακριβώς λόγω της κρίσης των ακινήτων. Ε, Επίση τι γίνεται με του άστεγους. Ζουν στον δρόμο, οι άλλοι δεν έχουν σπίτι και για κάποιο διάστημα μένουν με άλλους και κάποιοι άλλοι φιλοξενούν πρόσφυγες διότι δεν θέλουν να είναι ε, σε κάποιο χώρο, σε κάποια δομή κρατική οπότε έχουν, αυτοί, αυτοί αναγκάζονται να φιλοξενήσουν κάποιον που δεν έχει σπίτι όχι αναγκαστικά κάποιον που ζει στο δρόμο, αλλά και αυτοί είναι άνθρωποι ε, άστεγοι τελικά, μια που δεν έχουν στέγη. Επίσης, εγώ είμαι συμπρόεδρος του Intergroup για τους ΛΟΑΔΚΙ και με ενδιαφέρει αυτό που είπατε για τα ζευγάρια του ίδιου φίλου. Τι γίνεται στις χώρες που έχει νομιμοποιηθεί ο γάμος τέτοιων ζευγαριών. Ποια διαφορά υπάρχει σχέση με τις άλλες. Α, επίσης, λέει ο κύριος Άντζελ, είπατε ότι αυτοί που έχουν παιδιά δουλεύουν περισσότερο αυτούς που δεν έχουν. Αυτό πώς αναλύεται. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Και η Πρόεδρος λέει... Συμφωνώ, ήθελα εγώ και να το ρωτήσω το ίδιο. Μας δώσατε κάποια στοιχεία και μας είπατε επίσης ότι το 1 των ε, νοικοκυριών είναι οικογένειες μονοπρόσωπες. Τι, τι ισχύει αυτό για νέους ή για πιο ηλικιωμένους. Θυμάμαι επίσης ότι όταν ε, μετακόμισα για να σπουδάσω ε, συγκατοίκησα με άλλους γιατί ήταν πολύ ακριβά τα νίκια. Ε, αυτό κάνουν οι φοιτητές. Για πέστε μας, αυτό αποτυπώνεται στην ε, μελέτη. Επίσης, τι γίνεται για τις οικογένειες από ένα ζευγάρι, ιδίου ή διαφορετικού φίλου. Ε, τι γίνεται εκεί με ε, τα ζευγάρια χαμηλού εισοδήματο. Ε, αυτό ως μεταβλητή επηρεάζει το αν αποφασίζουν να κάνουν παιδί ή όχι. Ζητώ συγγνώμη, έχω και εγώ μια ερώτηση. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την πολύ πλήρη και αναλυτική έκθεσή σας. Στην ουσία όμως η έκθεση αυτή παρουσιάζει γνωστά θέματα. Εγώ αυτό που ε, ήθελα να ακούσω ήταν ο ορισμός της οικογένειας, διότι στις ε, διάφορες χώρες έχει, ορίζεται διαφορετικά. Ε, εμείς λέμε ότι όπου υπάρχει παιδί υπάρχει οικογένεια έτσι να συμπεριλαμβάνονται και τα ομόφυλα ζευγάρια ή οι παππούδες που αναθρέφουν ένα παιδί. Αλλά ε, στα, στις άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικοί ορισμοί. Ε, χωρίς την οικογένεια δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Είπατε κι εσείς ε, στην έκθεσή σας ότι πρέπει να δημιουργήσουμε την, τις συνθήκες πλαίσιο για την φροντίδα των παιδιών ώστε οι μόνοι γονείς να μπορούν να να, να εργάζονται. Ε, άσχετα όμως από τον, την δυνατότητα εργασίας. Ε, είπατε ότι η γυναίκα κάνει τις περισσότερες οικιακές εργασίες ε, και οι κατάλληλες δομές θα μπορούσαν να επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναθρέφουν ε, τα παιδιά όπως τα θέλουν και όπως θέλουν και όχι να δαπανούμε δισεκατομμύρια σε δομές φροντίδας των παιδιών. Ε, πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε, αλλά ε, δεν μας αναφέρουν τις προοπτικές για το μέλλον. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ λέει η ομιλήτρια, η κυρία Σαντόρ. Για να αρχίσουμε από τα νοικοκυριά χωρίς οικογένεια. Διαπιστώθηκε ότι είναι από άλλη χώρα οι νεότεροι. Όχι αναγκαστικά μετανάστες. κρίση σε όλη την σε όλη την Ευρώπη, αλλού ήταν χειρότερη κρίση όπως στην Ιρλανδία. Και επιστάσαμε ότι πάνε να μείνουμε με τους γονείς τους. Ε, ακριβώς λόγω της κρίσης των ακινήτων και της αύξησης των ενοικίων. Όχι, για τους άστεγους άλλοι ασχολήθηκαν. Καλά, θα κάνουμε άλλη έκθεση για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα για τα ομόφυλα ζευγαρία. Δεν καλύπτονται επαρκώς από τις επίσημες στατιστικές. Περισσότερα τέτοια ζευγάρια εκεί όπου έχει νομιμοποιηθεί ο γάμος τους. Περιορισμένα στοιχεία πάντως έχουμε για αυτά τα ζευγαριά, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε ανάλυση αναχώρα. Για τους πατέρες τώρα που δουλεύουν περισσότερο, ε, αυτοί θα πρέπει να καλύψουν την οικογένειά τους. Κυρίως εκείνοι που είχαν μεγαλύτερο εισόδημα το κάνουν αυτό. Πάντω, οι μητέρες δουλεύουν το ίδιο και στι δύο περιπτώσεις. Τώρα, τους μόνους γονείς και το χάσμα Ανατολής Δύσης. Σαν και Ευρώπη περισσότερο έντονο. Μόνοι, ηλικιωμένοι από όσο στη Δύση και ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία. Εκεί οι ε, οικογένειες με ένα μέλος είναι από νεότεροι άνθρωποι τέλο πάντων. Όπως είπαμε, ανά περιοχή έχουμε μεγάλες διαφορές. Ε, βέβαια και ο ορισμός οικογένεια διαφέρει από χώρα σε χώρα, οπότε και εμείς αποφύγουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες για τις διαστάσεις της κάθε οικογένειας. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη οικογένεια που δεν καλύπτονται, όπως κάποιοι που έχουν σχέση αλλά ζουν σε διαφορετικά σπίτια. Υπάρχουν επομένω νέα είδη οικογενειών. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα, περισσότερα στοιχεία για να εξετάσουμε καλύτερα το θέμα. Υπάρχουν εναλλακτικέ. Έχουμε και τους ε, παππούδες που φροντίζουν τα εγγόνια. Δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Και θα πρέπει να δούμε ότι δεν είναι πάντα αυτονόητο, δεν είναι εύκολο να έχουν εξωτερική βοήθεια οι γονείς για τα παιδιά τους. Οπότε επιστατεύουν τους παππούδες. Σε πολλές χώρες, ας πούμε στη Γερμανία, οι, οι μόνοι γονείς ζητούν τέτοια εξωτερική βοήθεια περισσότερο.